Good afternoon everyone. If you would like to take your seat, maybe... Καλησπέρα σα. Αν θέλετε να καθίσουμε για να ξεκινήσουμε. Πρώτο θέμα, η έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται χωρί τροποποίηση. Έχω να κάνω κάποιε ανακοινώσει. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την κοινή δημόσια ακρόαση επιτροπών Γιούρι και Έμβη για τις περιβαλλοντικές ευθύνες. Θα λάβει χώρα μια τέτοια ακρόαση για την εφαρμογή της οδηγίας περιβαλλοντικών ε, ευθυνών αύριο στις 3.30 το απόγευμα. Ε, ως τμήμα της ε, συνεδρίας της Επιτροπής Γιούρι. Υπάρχει μια έκθεση για την, μια διάμεση έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας ε, στην οποία η ΕΜΒΗ συμμετέχει γνωμοδοτούσα ε, και καλείστε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την αυριανή ακρόση. Δεύτερη ακρόση και δεύτερη ανακοίνωσή μου, ακρόση για την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το περιβάλλον, την ασφάλεια τροφίμων και της δημόσιας υγείας. 25 Απριλίου, Τρίτη 25 Απριλίου, η ημερομηνία της 4.30 το απόγευμα με συμμετοχή καλεσμένων ομιλητών όπως ο Τότ Στέρν, ο πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα, εκπροσώπους ε, του κλάδου, ε, των επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεων καταναλωτών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των ε, οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Καλείστε και εκεί να συμμετάσχετε. Για σήμερα έχουμε διαρμία σε 21 γλώσσες και ως συνήθως ε, ο φάκελος συνεδρίασης είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά ενώ η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ζωντανά. Έγκριση πρακτικών της 15ης Δεκεμβρίου, 12η Ιανουαρίου, 27η και 28 Φεβρουαρίου, καθώς επίσης και της 9 η Μαρτίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι τα ε, πρακτικά εγκρίνονται. Συστάσεις των συντονιστών της 21ης Μαρτίου. Διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξη. Σημείο 5. Η υποφαινόμενη θα σας ε, παρουσιάσει την, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου για το σύστημα εμπορίας εκπομπών πρώτη συνεδρίαση έγινε ήδη, βασίστηκε στις ε, βασικές θέσεις του Κοινοβουλίου ε, της 15 Φεβρουαρίου και στην γενική προσέγγιση του Συμβουλίου της 28 Φεβρουαρίου ε, που δεν προσαρμόστηκε με βάση τις δικητατικά μας σχόλια. Το Κοινοβούλιο του συμβουλίου και η Κομισιόν έκαναν μια ανταλλαγή απόψεων για τα πιο σημαντικά πολιτικά θέματα. Ορισμένες ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο, κοινο, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υπογραμμίστηκαν και ζητήθηκε να γίνει η εργασία σε τεχνικό επίπεδο σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα καλύτερη ε, προσαρμογή στα επίπεδα παραγωγής, τα benchmarks, οι μικροί ε, εκπέμποντες, η απλοποίηση, η ποιοτική αξιολόγηση, η έκθεση για, τον, για την αγορά άνθρακα, η αναθεώρηση του Παρισιού, το Ταμείο Καινοτομία και η Ελλάδα. Ο ζήτησα να, γίνει μία ακόμα συνεδρίαση υπό την Μαλτέζικη Προεδρία και ο πρόεδρος συμφώνησε. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται εκ των υστέρων από ό,τι φάνηκε δεν υπάρχει χώρος και ίσως διάθεση για μια πρόσθετη συνεδρίαση. Οπότε θα παραμείνουμε στο πρόγραμμα όπως είχε. Τεχνικές συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα πριν την επόμενη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου. Αν οι εμπειρογνώμονες εντοπίσουν θέματα τα οποία είναι πολιτικής φύσεως, τότε θα μας αναπέμψουν τη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα των τεχνικών συναντήσεων θα υποβληθούν στις διαπραγματευτικές ομάδες προκειμένου να συμφωνηθούν. Αυτά σε ό,τι αφορά την έκθεσή μου για τα πεπραγμένα. Επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ακρόαση της υποψήφιας ε, για την θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πλόρυψη, ε, και Ελέγχου Νόσων του ECDC. Η κυρία μου είναι μαζί μας, έχει προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ECDC 22 Μαρτίου για τη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Όπως προβλέπεται από την νομοθεσία που διέπει το ECDC, πριν διοριστεί, καλείται να απευθυνθεί στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα τις υποβάλουν τα μέλη. Η κυρία μου ε, είναι γνωστή μας διότι ε, την είχαμε, είχαμε ανταλλάξει μαζί τις απόψεις σε μια προηγούμενη φάση όταν ήταν προσωρινή ε, διευθύντρια του ECDC στις 15 Μαΐου. Γνωρίζουμε ότι ξέρει, ε, από, ξέρει τα θέματα του ECDC. Πριν την ακούσουμε να σας ενημερώσω για τη διαδικασία. Καταρχήν η κυρία Αμό ε, θα έχει στη διάθεσή της το πολύ 10 λεπτά για μια εισαγωγική τοποθέτηση. Μετά θα έχουμε ερωτήσεις από τους συντονιστές ε, ή τους αντιπροσώπους τους. 5 λεπτά ο καθένας. Μια, ένα λεπτό η ερώτηση για ένα θέμα, παρακαλώ, ένα λεπτό για ένα θέμα, όχι πέντε θέματα σε ένα λεπτό, γιατί δεν θα μπορέσει να τα απαντήσει η κυρία μου. Μετά θα δώσουμε στην κυρία μου δύο λεπτά να απαντήσει και μετά μια ανταπάντηση, ενδεχομένως 45 δευτερολέπτων με μια ε, συναφή ερώτηση και ένα λεπτό στην κυρία μου για να απαντήσει στην δεύτερη αυτή συναφή ερώτηση. Στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων θα έχουμε 12 ερωτήσεις από βουλευτές σε μπλοκ των τριών λεπτών δεν θα έχουμε ανταπαντήσεις ή ε, ε, δεύτερες ερωτήσεις. Και τέλος θα δώσουμε και πέντε λεπτά το πολύ στην κυρία μου για να κλείσει την ακρόαση αυτή με μια τοποθετησία. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair, members of the Committee. It's an honor and a pleasure to be here today. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή εμένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Τα χρόνια ήμουν η διευθύντρια, εκτελούσα αυτή διευθύντριας ε, για το ECDC και εξελέγην στην θέση αυτή τα τελευταία δύο χρόνια. Είχα πολλές ε, ευκαιρίες και δυνατότητες να συζητήσω μαζί σας για το πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τη στρατηγική μας ε, για το κέντρο. Θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιάσω τις ε, επιτυχίες μου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Είμαι γιατρός με πτυχίο για θέματα δημόσιας υγείας στη Γερμανία. Ξεκίνησα πριν από 20 χρόνια σαν μέρος του προγράμματος ΕΒΕΤ. Ήδη από τότε αλλά και μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αυτό είχε σαν σκοπό να περιορίσει την επέκταση των λιμωδών νοσημάτων στην Ευρώπη, κάνοντας μελέτες επιδημολογικές και βεβαίως είχε αποστολές ε, παρόμοιες με αυτές του ECDC. Ήμουν για τα τελευταία χρόνια μέλος της ομάδας που είχε σαν ε, κύρια αποστολή τον περιορισμό της επέκτασης αυτών των νοσημάτων, καθώς και τα έκτακτα περιστατικά. Ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο αναπτύξαμε και υλοποίησαμε, ιδιαίτερα για τα τελευταία χρόνια. Ήδη από το Μάιο του 2015 ήμουν επικεφαλής ε, τα προηγούμενα χρόνια του οργανισμού του ερευνητικού και βεβαίως ε, από την στιγμή που ανέλαβα έχω αναλάβει και καθήκοντα διοικητικά, κάτι το οποίο θα συνεχίσω για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πριν μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την αποστολή μου στο ECDC, θα ήθελα να περιγράψω την κατάσταση In Europe we see an increased στην οποία βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι ο ευρωσκεπτικισμός, ο οποίος ε, διαρκώς ε, επεκτείνεται στην Ευρώπη, το Brexit που είναι σήμερα μια πραγματικότητα, τα θέματα της ασφάλειας και ο, η αμφισβήτηση της ε, επιστήμης είναι κάτι που βεβαίως και αυξάνει την πίεση για όλους τους επιστήμονες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα τα δημογραφικά, η γεννητικότητα μειώνεται, οι μεταναστευτικές ροές και οι τεχνολογίες, οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε θέματα δημόσιας υγείας, ηλεκτρονική αν θέλετε, αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων δημόσιας υγείας, ε, καθώς ε, και το θέματα που αφορούν το DNA. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να πούμε ποια είναι η χρυσή τομή μεταξύ των διαφόρων μέσων αντιμετώπισης προβλημάτων ε, δημόσιας υγείας. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν τρόποι για να προβλέψει κανείς συγκεκριμένες ασθένειες μέσω εμβολιασμού η συνεχής επαγρύπνηση για την μη επέκταση γνωστών ασθενειών όπως ε, το AIDS, ο περιορισμός ε, του ιού ε, HIV, η νέα χρήση εμβολίων, η καλύτερη χρήση των εμβολιασμών, Όλα αυτά με σκοπό να υλοποιήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2020 των Ηνωμένων Εθνών η υπατήτηδα, η φυματίωση αλλά και το σιός HIV παραμένουν προτεραιότητες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπαγρυπνούμε. Υπάρχουν και νέε απειλές προς τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει λοιπόν το ECDC να συνεχίσει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε κρίση για τις ε, λοιμώδεις, που αφορούν τις λοιμώδεις ασθένειες. Είναι θέματα που σαφώς αφορούν και την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτές ε, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που έχουν την καλύτερη αποτελεσματικότητα, εντοπίζοντας προτεραιότητες με όλα τα συμβαλώμενα μέρη. Πρέπει σήμερα να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους, αποτιμημένους και με τον ίδιο τρόπο που εμπλέξαμε μέχρι σήμερα όλα τα συμβαλόμενα μέρη, να εντοπίσουμε και να συγκεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας στις στρατηγικές αυτές που αποφεύγουν τις επικαλύψεις και αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας. Θέλω να βελτιώσω την οργάνωση, θέλω να βελτιώσω τις σημερινές στρατηγικές, με κάθε τρόπο να βελτιώσω τις σημερινές στρατηγικές έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ε, υπεραξία του ECDC, την προστιθέμενη αξία, την αποτελεσματικότητά μας κατά νέων ασθενειών, νέων απειλών. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε κοινή δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Θα πρέπει να στηριχθούμε σε όλους τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δίκτυα αποτελεσματικά έτσι ώστε να μπορέσει το κέντρο μας να παίξει το, ένα καθοριστικό ρόλο. Θα ήθελα επίσης να συνεχίσω με τις συνεργασίες που είχαμε μέχρι τώρα και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με εσά που είστε τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα ήθελα επίσης να ενισχύσω τη συνεργασία που έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε με την ΕΦΣΑ και με όλες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, υπηρεσία φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι γνωρίζουμε ότι στις γειτονικές χώρες, στις τρίτες χώρες, υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν οι εταιρικέ σχέσεις. Το ΙΣΔΙΣΗ ήδη σήμερα έχει πολύ καλές συνεργασίες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τα κέντρα πρόβλεψης παντού στον κόσμο, με την παρακολούθηση των ασθενειών. Είναι κάποιες συνεργασίες και εταιρικέ σχέσεις που πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε στο μέλλον. Επισκέφτηκα το Αφρικανικό Κέντρο Πρόληψης των ε, Ασθενειών. Εκεί βεβαίως γνωρίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Μέχρι το 2022 έχω συγκεκριμένους στόχους. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κέντρο να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τις ε, εμπειρογνωμοσύνες, για τις συμβουλές που παρέχουμε. Για μένα ο κύριος στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτές τις στρατηγικές. Μέχρι τώρα η εργασία μας θα πρέπει να αποτιμηθεί και να βελτιωθεί. Είμαστε ένας εταίρος άλλων οργανισμών που συνεργάζονται παντού στον κόσμο για την προστασία όλων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ίση αντιμετώπιση όλων των ασθενειών και ίση προστασία όλων των κατηγοριών και των ομάδων. Πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βελτιώσουμε και τα εργαλεία πρόληψης. Τα έργα, οι μελέτες που έχουν αρχίσει θα πρέπει να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για τους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Επεγρυπνούμε επίσης έτσι ώστε να υπάρχουν σωστά κίνητρα για όλους όσους εργάζονται στο ECDC. Ολοκληρώνω την ε, μελέτη μου, υπενθυμίζοντα ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είμαστε αλλαζόνες, γιατί όλοι μας η δράση στο παρελθόν θα πρέπει να μας χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Εγώ, σαν διευθύντρια του ECDC, θα ήθελα να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα παίξει να παίξουμε στην παγίδα αυτή που μας περιέγραψε ο William Pollard. Ευχαριστούμε την παρουσία σα. Κύριε Αμών, και τώρα ερωτήσει και από του συντονιστέ. Σα υπενθυμίζω ότι έχουν ένα λεπτό για την ε, ερώτηση, άρα μείνετε σε ένα θέμα να ερώτηση. Πρώτος βέβαια ο κύριος Λίζε για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ πολύ την κυρία Χάμον. Χαίρομαι που βρέθηκε λύση, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε έναν ε, λεγμένο πρόεδρο, επίσημο πρόεδρο του ACDC. Συγκεκριμένα λοιπόν, η ερώτησή μου είναι για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Συγκεκριμένα, τι σχέδιο έχετε και τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου έχουμε πολλές φορές ε, υποβάλει προτάσεις για το θέμα αυτό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατή πρόταση νομοθετική από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς είμαστε κάπως αδύναμα εκπροσωπημένοι εδώ στην ε, αίθουσα αυτή σήμερα και ο Καν Μπόιλς ο οποίος ε, θα μπορούσε, αν ήταν εδώ, να σας έκανε πολύ πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις από μένα. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θα είναι η απόφασή σας για τα θέματα αυτά που ακόμη εκκρεμούν και για τα οποία δεν έχετε τόσο καιρό ε, δώσει καμία απάντηση. Συγκεκριμένα για το EMR. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο είναι ένα σχέδιο δράσης ε, για το θέμα της αντίστασης. Εμείς συνεισφέρουμε σε αυτό με τα στοιχεία που διαθέτουμε, τα δεδομένα που διαθέτουμε, την αξιολόγηση του κινδύνου και οτιδήποτε άλλο εμπεριέχεται στη στρατηγική για την αντιμετώπιση των ε, λοιμόξεων και τον έλεγχο των λοιμόξεων. Βεβαίως εμείς είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής για να μπορέσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε όσο μας το επιτρέπει η δική μας εντολή. Αν παραδείγματο χάρη χρειάζονται αποδείξεις, μετρήσεις, ε, ε, επιστημονικά στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσει να είναι αποτελεσματική η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση όσον αφορά την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Το θέμα της, ε, του αρισμού μιας ημέρας ε, για την συνειδητοποίηση της δράσης ε, των αντιβιωτικών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει επικοινωνία, να υπάρξει συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τους δώσουμε στοιχεία, δεδομένα, μηνύματα, λέγοντας ότι θα πρέπει όλοι να βασιστούμε σε κοινά μηνύματα, σε κοινή ενημέρωση και όλοι να πάρουν το ίδιο μήνυμα. Χρειάζεται επίσης να εργαστούμε και με τις χώρες ξεχωριστά είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε το μήνυμα στα δεδομένα της κάθε χώρας έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό, για να γίνει δεκτό. Και αυτό βεβαίως όχι μόνο για το θέμα του ΕΜΑΡ e αλλά και για άλλους τομείς. Για τη δεύτερη ερώτηση, όμως, θα μπορούσατε να απαντήσετε γιατί εγώ δεν μίλησα μόνο και για τα αντιβιωτικά, αλλά για την εργασία στο SDC γενικότερα. Δηλαδή, τι γενικότερα θα μπορούσατε να κάνετε έτσι ώστε να συνεισφέρετε στην σωστή λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που να περνούν αποτελεσματικά, να γίνονται κατανοητές ε, και εύληπτες από τους Ευρωπαίους πολίτες και να υπάρχει και περισσότερη διαφάνεια. Uh, αυτό δεν ήταν ουσιαστικά ερώτηση, αλλά συμφωνώ. Γι' αυτό σας ε, ανέφερα αυτές τις ε, ημέρες αφιερωμένες στα, στη χρήση των αντιβιωτικών, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να αγγίξουμε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό κάνουμε τώρα. Το κάνουμε αυτό για ε, τα εμβόλια. Ε, θα πρέπει βέβαια κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα της χώρας. Και βέβαια εσείς που ξέρετε καλύτερα την εκλογική σας περιφέρεια, αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε και έτσι να εφαρμόζεται κάθε φορά αυτή η υπόθεση στις ιδιορυθμίες της χώρας. Κύριε Αντάλιν, η επόμενη για τους σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ήρθατε και πάλι δόκτωρα Αμών. Χαιρόμαστε που σας ξαναέχουμε να ξανασυζητήσουμε για τόσο σημαντικά ζητήματα για όλο τον κόσμο στην πατρίδα μας τότε που εκτελούσατε καθήκοντα διευθυντή, ήταν μια περίπτωση δύο τόνων όπου αποδείξατε τι μπορείτε να κάνετε. Και εμείς ελπίζουμε ότι σε αυτή τη ρότα θα συνεχίσετε. Έχω κάτι να σας ρωτήσω που ανισχύει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ένωση σήμερα. Είπαν ότι σε 11 κράτη-μέλη, αλλά και στη Ρουμανία υπάρχει αυτή η επιδημία μόνο στην Ρουμανία 3.000. Πρόκειται για μαγουλάδες. Είναι μολυσματική ασθένεια και κανείς δεν προστατεύεται επομένω από αυτού του είδους ε, την επιδημία. Είναι κάτι επομένω το οποίο αφορά όλα τα κράτη-μέλη, γιατί αφορά επίσης και τα παιδιά. Η υπηρεσία σα, τι μπορεί να κάνει για να συγκρατήσει αυτό το φαινόμενο, αυτή την επιδημία. Κύριε Αμών, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ο είναι βέβαια ένα παράδειγμα κατά το οποίο Α, έχουμε τώρα αυτή την επιδημία που έχει ξεσπάσει σε 11 χώρες και περισσότερο έχει πληγεί η Ρουμανία. Αλλά θεωρούμε ότι είναι ενδεικτική περίπτωση. Φαίνεται τι γίνεται όταν δεν χρησιμοποιούμε εμβόλια όσο θα μπορούσαμε και όσο θα έπρεπε. Και δεν θέλω να κατηγορήσω καμία χώρα, Η Ρουμανία, ξέρετε, σε πρώτες είναι κάτω από τα τέσσερα έτη ο και στο Βέλγιο οι περισσότεροι είναι πάνω από 15 που έχουν χτυπηθεί και επομένως βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε κάθε φορά ποιος είναι ο πληθυσμός ο πιο ευάλωτος που τίνει να αρρωστήσει γιατί μπορούμε έτσι να τους καλύψουμε. Και έτσι επίσης έχουμε καλύτερα στοιχεία. Και έτσι μπορεί να είναι πιο καλά στοχευμένα τα μέτρα. Αυτό χρειάζεται. Καταρχήν τα πράγματα είναι απλά. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση, μην υπάρχουν κενά και να δούμε τι γίνεται με τη μετάδοση την αλυσίδα της μετάδοσης, να δούμε υπό ποιες συνθήκες ε, ζουν, βρίσκονται οι ασθενείς και έτσι προχωρούμε. Καταρχήν είναι πολύ απλό. Βάλει. Μα ακριβώ αυτό μας είπατε στην αρχή. Μας είπατε για τις επιφυλάξεις, αυτόν τον σκεπτικισμό όσον αφορά ε, το, το δισταγμό του κόσμου να προσφύγει στα εμβόλια. Πρόκειται για ηλαρά διορθώνει δερμηνία. Οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν το να κάνει ο κόσμο το εμβολίο και έτσι να μπορέσουμε να εκριζώσουμε το φαινόμενο αυτό τη ηλαρά στην Ένωση. Ναι, λέει κύριε Μόν, ε, έχουμε κάποιο είδου εργαλεία επικοινωνία για του εργαζόμενου στον τομέα τη υγεία και έτσι να μπορέσουμε να χειριστούμε ούτω ή του γονεί, να του καλύψουμε για ό,τι πρόβλημα έχουν, ό,τι ερώτηση έχουν να μας κάνουν για το πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια. Αυτό ακριβώς σας είπα και προηγουμένως. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στο τι ισχύει σε κάθε χώρα. Ίσως θα πρέπει αλλιώς να έρχομαστε σε επαφή με όσους έχουν μικρά παιδιά από ότι με όσους έχουν ε, έφηβους, αλλά τόσο πάντων έτσι θα πρέπει να δουλέψουν σε κάθε χώρα. Τώρα κατευθυντήριες υπάρχουν. Απλώς θα πρέπει κάποιος να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Βαλέαν. Ευχαριστώ. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Δόκτωρα Μον, που είσαστε μαζί μας σήμερα. Με χαρά θα δούμε ξανά ένα πραγματικό εκτελεστικό διευθυντή μετά από αρκετά χρόνια στον ECDC. Όπως είπε και ο κύριος ε, Λίζε, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στην, ε, μικροβιακή αντίσταση, στην αντιμικροβιακή αντίσταση. Η απογράφηση της Κομισιόν έληξε πέρσι, οπότε χρειαζόμαστε καινούρια μέτρα. Ερώτηση λοιπόν είναι, πιστεύετε κι εσείς ότι χρειάζεται πιο δραστήρια, ένα πιο δραστήριο, ε, πιο δραστικό πρόγραμμα εργασίας από τα περισμένα χρόνια. Και έχοντας υπόψη και την ε, απάντηση που δώσατε στον Πίτερ Λίζε, να σας ρωτήσω το εξής. Ε, ποια είναι η άποψή σας για τη διεθνή συνεργασία. Δείξατε το χάρτη που περιλαμβάνει και τους Κινέζους και κλπ. Ξέρουμε ότι ε, τα, σούπερ, τα υπερμικρόβια και οι υπερβραβεροί οργανισμοί εξαπλώνονται παντού σε όλο τον κόσμο. Μπορεί εμείς εδώ να είμαστε μια χαρά, αλλά χωρίς τη διεθνή Συνασία τι μπορούμε να καταφέρουμε. Απάντηση. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δράση Είχαμε πρόγραμμα δράσης και, και η Κομισιόν το είχε αξιολογήσει μάλιστα αξιολόγησε το αποτέλεσμα. Αυτή η αξιολόγηση έδειξε ότι πετύχαμε αρκετά πράγματα αλλά υπολοιπόμαστε του βέλτιστου. Και εκεί μπορούμε να δούμε το πρόγραμμα δράσης ε, σε συνδυασμό με αύξηση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Πολύ σωστά είπατε ότι το πρόβλημα αυτό είναι παγκόσμιο. Ελπίζουμε ότι η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τις σημαντικές μεγάλες χώρες του κόσμου θα μας βοηθήσει να απαντήσουν, να δώσουμε μία απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε την συνεργασία TATFAR με τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Ήδη από, εκεί από τότε προσπαθήσαμε να συντονίσουμε τις εργασίες μας. Παρ' όλα αυτά, κατά την άποψή μου, μπορούμε να ε, επικεντρώσουμε και να κάνουμε πιο ισχυρή τη συνεργασία μας με πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα την Ινδία. Γιατί από την Ινδία έρχονται στελέχη που πραγματικά ανθίστανται στα αντιβιωτικά πολύ. Ε, κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω την δόκτωρα Μον γιατί στις δύσκολες στιγμές που ο ECDC δεν είχε ένα μόνιμο εκτελεστικό διευθυντή ανέλαβε τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή και έκανε εξαιρετική δουλειά. Τα στελέχη του ECDC νομίζω ότι ε, την εκτίμησαν ιδιαίτερα, οργάνωσε πολύ καλύτερα τον οργανισμό, προετοίμασε τα γραφεία στα οποία θα μετακινηθεί του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνατε στον ECDC, κυρία μου, δόκτωρα μου. Κάποιοι που δεν πρόσεχαν πολύ κοντά το τι συνέβαινε, Ενδεχομένω δεν θα είχαν καταλάβει καν ότι υφίστατο κάποια απουσία ε, στο οργανόγραμμα. Μιλήσατε για τη συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις και οργανισμούς. Σίγουρα δεν μπορεί ο καθένας να είναι μοναχικός καβαλάρης. Θα μπορούσατε όμως να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς φαντάζεστε με την συνεργασία, για παράδειγμα με την EMA. Ευχαριστώ. Yeah, I mean we... Απάντηση. Ήδη συνεργαζόμαστε με την EMA. Για παράδειγμα, σε θέματα αντιμικροβιακής αντίστασης ε, και εμβολιασμών. Προσπαθούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες με τον EMA προκειμένου να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Ένα παράδειγμα είναι η κοινή μας έκθεση για την αντιμικροβιακή ε, αντίσταση σε ζώα και σε ανθρώπους. Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2015 και μια δεύτερη εκδοσή θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Θέλουμε οι ειδικοί να έχουν πλήρη εικόνα με βάση τα στοιχεία που έχουμε και εμείς και ο EMA. Με τον EMA ε, επίσης συνεργαζόμαστε σε θέματα εμβολιασμών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τροφίμων εξετάζει την ασφάλεια των εμβολιασμών, εμείς την αποτελεσματικότητα, οπότε εκεί αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό που επίσης θέλω να αναπτύξω με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς είναι όχι μόνο να ανταλλάσσουμε πρόγραμματα εργασία όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά όταν προγραμματίζουμε τις μελλοντικές μα εργασίες, να το συζητάμε μεταξύ μας. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ε, σύνταξης της επεξεργασίας των ε, προγραμμάτων εργασίας μας, να συζητούμε. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Σας ρωτώ, διαπιστώνετε επίσης να υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε σχέση με το πλαίσιο που έχετε θέσει μέχρι τώρα. Τι μπορεί να γίνει στις μολυσματικές ασθένειες περισσότερο, τι μπορεί να γίνει από νομοθετικής πλευρά στην Ευρώπη. ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει λόγος να ενεργεί. Κοιτάξτε τι εννοείται, εννοείται να διευρύνουμε την εντολή μας για τις μολυσματικές θένες περισσότερο ή να πάμε και σε άλλου είδους φαινόμενα πέραν των μολυσματικών μεταδοτικών. Ναι, ναι, ναι, για αυτές τις ασθένειες νομίζω ότι έχουμε τον κανονισμό που μας παρέχει ό,τι βάση χρειάζεται. Υπάρχει η εντολή για την αξιολόγηση κινδύνου, για να υπάρξει καθοδήγηση για τις επιλογές που υπάρχουν, τα μέτρα ελέγχου, αρμοδιότητα εθνική, αρμοδιότητα ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ναι, νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουμε εμείς κάποιες από εκείνες αρμοδιότητες. Ευχαρίστω να εργαστούμε τους συναδέλφους σε Επιτροπή και σε κρατημέλη. Τους παρέχουμε ό,τι στοιχεία υπάρχουν, ό,τι μέσα έχουμε, ούτως ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στα αναγκαία μέτρα για να πολεμήσουν τις κρίσεις που ξεσπούν τις ασθένειες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις ερωτήσεις που θα δώσετε. Όσον αφορά την ανταλλαγή ερωτήσεων, απαντήσεων και οι απαντήσει μα έχετε δώσει μέχρι τώρα την εμπειρία που έχετε όσον αφορά τι λοιμώδει ασθένειε. Βεβαίω, βλέπουμε ότι η προτεραιότητα της Προεδρίας της Μάλτας είναι αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία νόσων, οι μη μεταδοτικές, ε, καθότι έχουν πάρα πολλά θύματα. Βεβαίως υπάρχουν και κατηγορίες ε, λιμωδών νοσημάτων που βλέπουμε ότι έχουν επανέλθει και προκαλούν όλο και περισσότερες λοιμώξεις. Η κάλυψη από τον εμβολιαρισμό βλέπουμε να μειώνεται στην Ευρώπη. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι εξής. Με ποιο τρόπο θέλετε να ενισχύσετε τα προγράμματα παρακολούθησης των λοιμωδών νοσημάτων και τι ακριβώς θα κάνετε για να υπάρξει η βέλτιστη κάλυψη και εμβολιασμό σε περιοχές, ιδιαίτερα όταν γνωρίζει σήμερα κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα, παρενέργειες κάποιων τέτοιων εμβολίων και πολλές φορές ε, έλλειψη των συγκεκριμένων φαρμάκων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την παρακολούθηση για τις μεταδοτικές ασθένειες. Αυτό είναι κάτι που ήδη το επεξεργαζόμαστε στην στρατηγική μας με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε πολύ συγκεκριμένα να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα, όπως παραδείγματος χάρη, να διευκολύνουμε την μετάδοση πληροφοριών από μέρος των κρατών μελών. Φαίνεται ότι σήμερα υπάρχει δυσκολία και την ίδια ώρα θέλουμε τα στοιχεία που διαθέτουμε εμείς στο κέντρο παρακολούθησης να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από μέρους των κρατών μελών. Να γνωρίζει δηλαδή το κράτος μέλος τι ακριβώς υπάρχει στα δικά μας δεδομένα, ενώ γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση η οποία ισχύει στη χώρα τους να προετοιμάζουμε επίσης την αντιμετώπιση, την ε, αντιμετώπιση κάποιων συγκεκριμένων ασθενειών με κατάρτιση. Στηρίζουμε παραδείγματος χάρη την κατάρτιση στις χώρες. Στηρίζουμε όμως και την ανείχνευση κάποιων ε, ασθενειών από μέρους των εργαστηρίων που βρίσκονται στην κάθε χώρα. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα βεβαίως και ο εμβολιασμός και όλες οι πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε για να σταματήσουμε τη μετάδοση κάποιων ασθενειών. Η καταπολέμηση όσον αφορά τις ε, παρενέργειες των εμβολίων και ε, συγκεκριμένα η λανθασμένες ε, πληροφορίες για παρενέργειες εμβολίων. Βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τις ε, παρενέργειες ε, για κάποια εμβόλια, οι οποίες δεν είναι σωστές. Κάνατε και μία ερώτηση για την έλλειψη κάποιων φαρμάκων και κάποιων εμβολίων. Βεβαίως και θα πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ελλείψεις αυτές με μεταφορά από τη μια χώρα στην άλλη παραδείγματος χάρη. Η κυρία Ντογνάνο, όταν σας μίλησα για κάποιες επισφαλείς ομάδες του πληθυσμού, εκεί ε, αναφερόμουν συγκεκριμένα στη φυματίωση, στην αντίσταση σε κάποια φάρμακα και ιδιαίτερα για άτομα που, έχουν, ε, που είναι φορείς του ιού HIV. Το εμβόλιο βάλων και βάλων για τα οποία στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη, πέρα δηλαδή από τα συνήθεια εμβόλια κατά της ε, διφθερίτιδας και του τετάνου. Θα ήθελα να μου πείτε ποια, κατά την άποψή σας, πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Ναι, όσον αφορά τις επισφαλείς ομάδες πληθυσμού, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ρωτάτε. Βεβαίως υπάρχουν πιο ευάλωτες κατηγορίες και ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από δύο από αυτές τις ασθένειες. Παραδείγματος χάρη τη φυματίωση και τον ιό του AIDS. Αυτές οι κατηγορίες θα πρέπει να εντοπίζονται στην κάθε χώρα και να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόληψη, πρόσβαση σε αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού και αυτό βεβαίως σε κάθε χώρα. Τώρα για τις ελλείψεις κάποιων εμβολίων, η πιο άμεση απάντησή μου και η πιο άμεση στήριξη που μπορούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη είναι μια καθοδήγηση για το πού υπάρχουν εμβόλια και πώς ε, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για κάποιους εμβολιασμούς. Αυτό είναι η πιο άμεση απάντηση που μπορούμε να έχουμε. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, Είτε θα πρέπει να υπάρχουν ανταλλαγές φαρμάκων και εμβολίων μεταξύ κρατών μελών, είτε κάποιες ε, κοινέ ε, αγορές, προμήθειες για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι και θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής που θα πρέπει σίγουρα να απασχολήσει και την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Το είναι ο και τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο. Λέει η πρόεδρος, έχουμε τώρα διαφορετικούς κανόνες. Ένα θέμα, ναι, ερώτηση και δεν υπάρχει επερώτηση στη συνέχεια. Ο πρώτο που θα υπόλοιπε ο κύριο Φαρία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία μου, δόκτωρα μου. Εγώ επισκέφθηκα τον CDC στην τελευταία μας επίσκεψη εκεί, ε, αποστολή εκεί και είδα πόσο καλά λειτουργεί. Η ερώτηση που απασχολεί πολλούς Πορτογάλους είναι η εξής. Γνωρίζετε ότι η πατήτηδα Α στην ε, Πορτογαλία έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο μεταξύ ανδρών ομοφιλοφίλων από τις άλλες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης. Πώς μπορεί ο ECDC ε να είναι πιο αποτελεσματικό στην ε, πανευρωπαϊκή ενημέρωση και έτσι ώστε τέτοιου είδους μεταδοτικές ασθένειες να εντοπίσουν και να περιορίζονται στα πρώτα του στάδια. Ευχαριστώ. Κυρία μου. Μιλάτε για την πατήτη Α, έτσι δεν είναι, ωραία. Η πατήτη Α είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν διότι υπάρχει έλλειψη εμβολίων. εξετάζουμε το ενδεχόμενο αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πατήτηδα Α αυτή τη στιγμή ε, είναι πολύ διαδομένη μεταξύ ομοφιλόφιλων ανδρών, ε, επηρεάζει δηλαδή μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί και στοχευμένα μέτρα πρόληψης. Η πρόληψη σίγουρα δεν μπορεί να γίνει μέσω ενός ανακοινοθέντος προς το γενικό πληθυσμό, προς την κοινή γνώμη στο σύνολό της. Πρέπει να διοχετεύσουμε το μήνυμα στα σωστά κανάλια. Στα κανάλια τα οποία φτάνουν στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Ε, έχουμε εμπειρία από τον ιό του AIDS και τη εργασία μας και τα ίδια κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ για την πατρίτιδα Α. Πάντως το σημαντικό είναι να γίνεται ο εμβολιασμός γιατί αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της πατρίδας Α. Συγχαρητήρια για τον διορισμό σας. Ε, συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει στον ECDC. Σας εύχομαι καλή πτυχία να συνεχίσετε εκεί που είσαστε. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε μιλήσει για τις μεταδοτικές ασθένειες και την αντιμικροβιακή ε, αντίσταση. Η ευρωπαϊκή δράση έχει εστιάσει στην ε, μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, όμως χαίρομαι που ε, ακούω ότι μιλάτε για μια στρατηγική ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε συνεργασία με το, τα κράτη-μέλη και την συγκεκριμένη πρόταση ε, εορτασμού μιας ημέρας ευαισθητοποίηση για το θέμα. Όμως μην ξεχνάμε και την έρευνα για εναλλακτικά φάρμακα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το ζήτημα και να ακούσω τη δική σας στρατηγική υποστήριξης της ε, έρευνας ε, εναλλακτικών φαρμάκων. Και κάτι πιο συγκεκριμένο. Ε, έχουμε έξαρση της πατήτητας Α και στη χώρα μου και στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν ξέρω αν έχετε μια ειδική στρατηγική για αυτό το θέμα. Okay. Uh, first question regard... Πρώτη ερώτηση, στρατηγική σχετικά με την έρευνα σε εναλλακτικά φάρμακα. Η έρευνα δεν εμπίπτει ακριβώς στο πεδίο μας. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το εξής. Αν υφίστανται εκθέσεις για αυτό το θέμα, να δούμε τι αποτελέσματα, επιστημονικά αποτελέσματα έχουν προκύψει για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένω. Ε, για να προωθήσουμε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία μόρια τα οποία έχουν ανακαλυφθεί. Εμείς δεν μπορούμε οι ίδιοι να κάνουμε κάτι στο επίπεδο της έρευνας. Σε ό,τι ιδέα αφορά την υπατήτη α, νομίζω ότι το είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι το μήνυμα θα πρέπει να περάσει στις κοινότητες των ομοφιλόφιλων ανδρών Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε καλύτερα αυτούς τους πληθυσμούς με προληπτικά μέτρα. Και βέβαια φαρμακευτική αγωγή αν υφίσταται. Eck. Κύριος Εκ είναι επόμενος. Ευχαριστώ. Κυρία Χάμον, Μιλήσαμε για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Έχουμε χιλιάδες ε, όμως θύματα και εκατοντάδες νεκρούς κάθε χρόνο. Και πιστεύω ότι και ο Επίτροπος Ανδρεοκάητης, ο οποίος έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό, αλλά εκφράστηκε λέγοντας ότι είναι μια πολύ σημαντική απειλή αυτή η αντίσταση σε πολλά αντιβιωτικά και συγκεκριμένα στα αντιβιωτικά λέγοντας ότι αυτή η απειλή διαρκώς ενισχύεται. Έχω την εντύπωση ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτή την απειλή και δεν συνειδητοποιούν ότι εμείς μιλάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψηφίζουμε για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, των ε, ε, σκυλιών, των μικρών ε, κατοικίδιων ζώων και δεν ε, αντιμετωπίζουμε σοβαρά το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα ότι πλέον πολλά μικρόβια, πολλοί ιοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη απειλή. Πρόκειται για μια απειλή που σήμερα όλο και περισσότερο απειλεί πολλές κατηγορίες ε, ζώων. Είναι ίσως καλύτερο σήμερα να κοιτάξουμε την ε, γεωργία, παραδείγματος χάρη, την ε, κτηνοτροφία. Ξέρουμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, ότι για τα κουνέλια υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία ζώων που δεν μπορούν να προστατευθούν και αυτό εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης αντιπιωτικών. Κοιτάξτε, εμάς η δική μας, αν θέλετε, αρμοδιότητα είναι η λοιμώδης νόση που απειλούν τους ανθρώπους. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα η προστασία κάποιων ζώων. Εκτός εάν υπάρχει μετάδοση από κάποιο ζώο σε έναν άνθρωπο, είτε πρόκειται για κτηνοτρόφο, είτε πρόκειται για κάποιον που φροντίζει αυτά τα ζώα. Η κατάσταση όσον αφορά τα ζώα δεν είναι καθόλου δική μας αρμοδιότητα και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που ήρθε για την κυρία Αμών. Εδώ και τρία χρόνια είμαι ευρωβουλευτής και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι έργο επιτελείται στο ECDC, γιατί είχαμε πολλές κρίσεις τις οποίες έχετε παρέμβει. Όμως θέλω κάτι να ρωτήσω σε σχέση με αυτό που ο κύριος Λίζα και ο κύριος Χερμπράντη. Τώρα τι κάνουμε. Για κοιτάξτε, τι ισχύουν με την, την μικροδιακή αντίσταση. Στις κάτω χώρες το θέμα ενδιαφέρει πολύ και εσείς μας μιλήσατε για ένα πρόγραμμα σχέδιο δράσης. Και ο κύριος Ανδριος είπε ότι θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της ασθένειας. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Θα μπορούσε να ασχοληθεί επ' αυτού και η Επιτροπή των Περιφερειών. Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που έρχονται να μας επισκεφτούν εδώ στη Βεξέλη και μητέρες που μας ε, λένε τα προβλήματά τους και ρωτάνε τι κάνουμε εμείς, τι κάνουν πολιτικές ομάδες, τι χρειάζεται κοινό με το παλιό δεν καταφέρνουμε τίποτα. Αλλιώς θα έχουμε απομόνωση. Ε, άρα χρειάζεται σχέδιο δράσης. Να εμπλακεί και η Επιτροπή των Περιφερειών και να δουλέψουμε με τον τύπο, τα ΜΜΕ, την τηλεόραση, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το πρόβλημα αυτό και την ε, αντιμικροβιακή αντίσταση. Για πέστε μας πώς το βλέπετε αυτό και τι πόροι οικονομικοί υπάρχουν σχετικά. Η κυρία Μόνο. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο θέμα Επιτροπής Περιφερειών, θα πρέπει όλοι να εμπλακούν. Επί μακροχρονικό διάστημα έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, προσπαθούμε να το προβάλλουμε, να ε, ενταχθεί στο θεματολόγιο των ηγετών Έγινε τελικά αυτό, το καταφέραμε και τώρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι όλοι χέρι-χέρι θα συντονιστούν, γιατί τίποτε δεν θα ήταν πιο επιζήμιο εάν ο καθένας έστελνε διαφορετικό μήνυμα στον κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο τώρα. Σας είπα προηγουμένως τι γίνεται όσον αφορά αυτή την μέρα συνειδητοποίησης τη ε, της των αντιβιωτικών είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι. Μη κυβερνητικέ οργανώσει, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ο ΠΟΗ που ασχολούνται. Και ο ΠΟΗ επίση καθιέρωσε μια εβδομάδα για την αντιπροεδρική αντίσταση, όπω και εμεί κάναμε αυτή την ημερίδα. Παράλληλα γίνεται αυτό τώρα. Το μήνυμα έχει ληφθεί από τις διάφορες χώρες, γίνονται σχετικές εκστρατείες ενημέρωσης εκεί που πρέπει. Φτάνουν τους γιατρούς, κάνουν τις συνταγές, ε, τα νοσοκομεία, αγγίζουν αυτές οι εκστρατείες, ε, γίνονται διάφορες παρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου, οπότε υπάρχει αυτή η πολλαπλή προσέγγιση που είπατε. Αυτό κάνουμε. Τώρα, αυτοί όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν προέρχονται μόνο από τον τομέα της δημοσίας υγείας, προέρχονται και από τον τομέα της φαραγωδιομηχανίας οι οδιοδοντίατροι, οι κτηνίατροι, άρα πρόκειται για ευρύ φάσμα κόσμου που προσπαθούμε να εμπλέξουμε και όλοι αυτοί επομένω έχουν εγγύψει το πρόβλημα. Υπάρχουν αποτελέσματα ή θα υπάρξουν, αλλά χρειάζεται υπομονή. Η κούρσα είναι μαραθώνιος. Ας περιμένουμε με ένα ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας για αποτελέσματα. Βαλεάν. Ευχαριστούμε. Κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια για το διορισμό σας και πιστεύω πραγματικά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική συνεργασία με τον οργανισμό τον οποίο προεδρεύεται. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως ε, τώρα σε μία άλλη υπηρεσία, στην ΕΦΣΑ. Ξέρετε βεβαίως ότι υπάρχει στενή συνεργασία και υπήρχε και στο παρελθόν μεταξύ ημών και τσέφσα. Μας έχουν απασχολήσει διάφορα θέματα, το θέμα της αλμονέλας, το πρόσφατο παρελθόν, το θέμα άλλων ε, βακτηρίων κάτι που θα θέλαμε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση με τον καταναλωτή και να υπάρχει καλύτερος τρόπος πρόληψη. Κοιτάξτε, η συνεργασία μεταξύ του ACDC και της ΕΦΣΑ είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζεται για κάθε είδους ασθένεια, απειλή που μπορεί να προέρχεται από τρόφιμα και τα οποία αφορά την ε, δημόσια υγεία. Έχουμε στοιχεία που αφορούν τα τρόφιμα, που αφορούν τα, τις ζωοτροφές και πρόκειται για μία έκθεση για τη δημόσια υγεία, δεν το ονομάζουμε έτσι, αλλά περί αυτού πρόκειται, που περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Και βεβαίως αυτό που κάνουμε μεταξύ του SDC και της ΕΦΣΑ δεν είναι απλώς κοινή ε, μελέτη, αλλά κάνουμε και κοινέ ε, ανακοινώσεις προς τον τύπο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κάποιες ε, επιδημίες, νέες επιδημίες και βεβαίως κάνουμε και αξιολόγηση του κινδύνου. Οι ομάδες μας συνεργάζονται, οι εμπειρογνώμονες της ΕΦΣΑ και του ECDC συνεργάζονται και προτείνουν κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαϊάκα. Ε, για τον HIV θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Γνωρίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει ε, διάγνωση νωρίς, ε, αυτό επιτρέπει τη λήψη αγωγής που μειώνει πολύ τις επιπλοκές. Ερώτηση λοιπόν είναι πώς, ποια είναι η δική σας στάση για αυτό το ζήτημα, δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Δεύτερον, τα τελευταία 30 χρόνια η επιστημονική πρόοδος ήταν σημαντική σε ό,τι αφορά ε, τον HIV. Τι συμπεράσματα μπορούν να βγουν από αυτό για άλλους τομείς της ανθρώπινης υγείας ε, και όμως και για το μέλλον της, ε, του, του HIV. Ε, Α ξεκινήσω από τον ιό του AIDS. Όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικό η διάγνωση να γίνει όσο πιο νωρίς είναι δυνατό. Και αυτοί οι οποίοι έχουν τον ιό να λάβουν την κατάλληλη αγωγή. Όμως, όταν δείτε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αυτοί αναφέρονται ειδικά στον HIV και ο στόχος είναι η ασθένεια να έχει εξαλειφθεί μέχρι το 2030. Όμως αυτή η προσέγγιση δεν πρόκειται να μας οδηγήσει στην επιτεύξη του στόχου. Για να πετύχουμε το στόχο του 2030 πρέπει να προχωρήσουμε πολύ και στην πρόληψη. Όχι μόνο στην ε, έγκαιρη διάγνωση. Και αυτό προσπαθούμε να προωθήσουμε πρόληψη. Προφανώς είναι πολύ καλό που διαθέτουμε πλέον φαρμακευτική αγωγή ε, που επιτρέπει στους ε, φορείς ε, να διάγουν μια σχεδόν κανονική φυσιολογική ζωή. Όμως θα είναι ακόμα καλύτερη η ζωή τους αν δεν είχαν τον HIV, θα ήταν καλύτερη. Γι' αυτό το λόγο από ηθικής, ιδεοντολογικής πλευράς αλλά και από οικονομικής πλευράς είναι καλύτερη πρόληψη. Αυτές οι αγωγές δεν είναι φτηνές. Καλύτερα λοιπόν η πρόληψη. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τα προεκτικά μας μέτρα. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με άλλες ασθένειες. Το κέντρο μας έχει ακριβώς τον τίτλο πρόληψης και ελέγχου των νόσων. Όχι μόνο ελέγχου, ε, αλλά και πρόληψης. Το αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν και με άλλες ασθένειες. Ευχαριστώ. Κυρία Ντάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πανέρχομαι, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε στα εισαγωγικά σας σχόλια. Θα επανέλθω σε κάποια από αυτά, γιατί είπατε με μεγάλη αποφασιστικότητα ότι πρέπει να ληφθεί άμεση ε, δράση και όχι μετά από ένα χρόνο. Καμιά φορά βέβαια είναι πιο εύκολο να το πει αυτό κανείς, ότι χρειάζεται άμεση δράση, αλλά η γραφειοκρατία και άλλα εμπόδια οδηγούν σε καθυστερήσεις και τελικά η αντίδραση, η δράση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση δράση και μάλλον θα έπρεπε να αντιδράσουμε χτες και όχι σήμερα. Πώς μπορείτε να προτείνεται κάποια επιτάχυνση της αντίδρασης, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ε, τέτοιου είδους περιπτώσεις που χρειάζονται άμεση δράση. Κοιτάξτε, αναφέρθηκα πιο συγκεκριμένα στην αξιολόγηση του κινδύνου. Γενικότερα όμως, ο εντοπισμός, ε, ο έγκαιρος εντοπισμός των απειλών Έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας έτσι ώστε οι διάφορες φήμες που κυκλοφορούν, οι πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επαληθευθεί να εξετάζονται πολύ νωρίς από μας για να μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια αξιόπιστη αξιολόγηση κινδύνου και να βασίσουμε την προληπτική μας δράση. Όχι μόνο την προληπτική μας δράση αλλά και τον έλεγχο κάποιων ε, ασθενειών. Πρέπει λοιπόν να υλοποιήσουμε άμεσα, να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα κάποιες επιδισμίες που μπορεί να ξεσπάσουν, κάποιες κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας ενισχύοντας τις δυνατότητες που διαθέτουμε, βελτιώνοντας τις δομές, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία κτλ. κτλ. Αυτό είναι για μένα μέρος της στρατηγικής μας με τις χώρες. Να στηρίξουμε δηλαδή, να βοηθήσουμε τις χώρες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα και πιο έγκαιρα όλα αυτά τα θέματα. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την ετοιμότητά μας και την δράση μας, βελτιώνοντας τη συνεργασία μας και ενισχύοντας τα κράτη-μέλη. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση θα είναι δική μου. Να σας ρωτήσω, λέει ο Πρόεδρος, ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα τα οποία έχετε από πλευράς της ε, υπηρεσίας, από πλευράς ε, προϋπολογισμού, από πλευράς ε, οικονομικών πόρων και τι μπορείτε να κάνετε ως ε, εκτελεστική διευθύντρια. Όπως σας είπα για τα προβλήματα που έχουν μπροστά μας, ναι υπάρχουν τέτοιου είδου οικονομικά ζητήματα τα οποία εντοπίζουμε και ε, τώρα για τις αρχές του επομένου έτους πρόκειται να ολοκληρώσουμε ε, αυτό το 10% για τις θέσεις που είχε αποφασιστεί το 2013. Οπότε θα έχουμε κάποιες άλλες περικοπές στους πόρους μας και κάποιες οροφές αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε επομένως εκεί που μπορούμε να ε, βγάλουμε ε, κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα. Θα πρέπει βέβαια πρώτα πρώτα να δούμε πώς θα είναι μετρήσιμη η επίπτωση της δράσης μας, γι' αυτό και είπαμε για δείκτες και για στόχους και επίσης θα πρέπει να υπάρχει διάλογος με τους ε, μπλεκομένους, να δούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες, που αποδίδουν περισσότερο. Άρα σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι πρεσβεύουν και εκείνοι, τι θεωρούν εκείνοι ότι είναι το πιο χρήσιμο. Αυτό εννοούσα όταν σας μίλησα σχετικά. Το πόσο είναι σημαντικό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα αποτελέσματα με τη δράση μας. Και αν κάτι βγει, θα είναι κάτι ποιοτικό, ανεξάρτητη φύση, αλλά τέλο πάντων, αν κανεί δεν το χρησιμοποιεί, τίποτα είναι χαμένα λεφτά. Άρα δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Να επικεντρωθούμε σε αυτά που είναι πιο χρήσιμα και να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά αυτά. Πάσε, σε ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για εσά, συνάδελφοι, για τι ερωτήσει σα και τώρα Κυρία μου, πρόκειται τώρα να δευτερολογήσει. Να κάνει μια σύνθεση των όσων ε, ρωτήσαμε, των όσων συζητήσαμε. Έχετε πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ για όλες σας τις ερωτήσεις, λέει η κυρία Μόν. Ίσως δεν τις απάντησα όσο εξαντλητικά θα θέλατε. Παρ' όλα αυτά, μου δείξατε και μου εκφράσατε τι για σας είναι σημαντικό. Ε, να είστε σίγουροι ότι αυτά θα ληφθούν υπόψη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς αυτό θα είναι η πηξίδα για να μπορέσουμε να βαδίσουμε στον πρώτο έργο μας τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς όπως περίμενα. Αυτά τα θέματα σας απασχολούν. Αυτά βλέπετε ως προτεραιότητα. Άλλωστε και τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε το πόσο θα πρέπει όλοι να έχουμε επίγνωση το ότι όλα όσα προγραμματίζουμε ακυρώνονται από κάποια κρίση που θα μπορούσε να σοβήσει. Μια πανδημία, μια γρήπη που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Οπότε, άρα όλα σε εκείνη την περίπτωση θα πρέπει να μπουν στο ψυγείο. Αυτό θέλω να σας επισημάνω. Ό,τι λέμε τώρα ίσως δεν ισχύσει για όλη τη διαδρομή. Ιδίω αυτό που είπατε στην τελευταία ερώτηση, που μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να σας επισημάνω ότι θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να δούμε τις αρνητικές προτεραιότητες. Δηλαδή, α, α, ακόμα και αν κάτι έχει επιπτώσεις, ακόμα και αν κάτι είναι αναγκαίο, μπορεί να μην μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί δεν θα έχουμε αρκετούς πόρους. Ακριβώς όπως είπαμε για την παγκόσμια συνεργασία. Μα και αυτή χρειάζεται πόρος. Θα πρέπει να βαδίσουμε με βάση τα όσα έχουμε. Και έτσι να δούμε τι επιλογές έχουμε να επεκτείνουμε το έργο μας. Ό,τι έχουμε, αν δεν έχουμε επιλογές, θα πρέπει να πάμε σε περικοπές. Γι' αυτό είπα ότι θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα ίσως από όσα τελικά θα καταφέρουμε. Βέβαια, και αυτό που είπαμε τελευταία φορά ήταν σημαντικό ότι όλες αυτές οι συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα και το τι βγαίνει, συμφωνώ, αλλά αυτό θα πρέπει να το αποσυνδέσουμε από τον στόχο μας, τον σκοπό μας δηλαδή, να αξιολογήσουμε, να εντοπίσουμε, να ενημερώσουμε για τις ασθένειες. Εάν μπορέσουμε να έχουμε επιπτώσεις από το έργο μας εκεί, τότε θα είμαστε χρήσιμοι μου. Οπότε, ακριβώς θέλω να σας πω ότι βάσει της εντολής μας θέλουμε την αποτελεσματικότητα στη δουλειά μας για τα θέματα που θεωρούμε σημαντικά. Εκεί να ενεργήσουμε όσο γίνεται με περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Αυτό θέλω να κάνουμε ως θεσμικό όργανο, ως οργανισμός. Και να αποσυρθούμε από άλλα μέτωπα που δεν είναι τόσο αναγκαία, που δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί. Αυτό θέλω να κάνω. ευχαριστώ, Αλλά δεν θέλω να υπονομεύσω τον σκοπό μας. Να έχουμε μόνο την προστέμινη αξία όσον αφορά τις ε, τα μεταδικές ασθενείς. Εδώ τελειώνουμε αυτή την ακρόαση με την υποψήφια για την, ε, το πόστο της εκτελεστικής διευθύντρες του ECDC συζήτηση θα γίνει στου ε, συντονιστέ και θα προετοιμάσουμε την έκθεσή μα για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάμπη. Now, dear colleagues, we move to... Περνάμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. Προσχέδιο έκθεσης του κυρίου Σεντάνς ε, για τους, τις δράσεις υπέρ των στόχων της ε, ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντάνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και τη στήριξή σας. Ε, πολύ καλή συνεργασία με τους άλλους και οδησηγητές και το προσωπικό τους το θέμα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης είναι τεράστιο και άπτεται σχεδόν όλων των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο λοιπόν ε, ένα πρόγραμμα δράσης να καλύπτει όλα τα πεδία τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Αυτό λοιπόν που ήθελα να κάνω και το υπογραμμίζω στην έκθεση είναι Ε, να μην θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς ένα κατάλογο με ένα checklist αλλά μια ολόκληρη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ θεσμικών οργάνων αλλά και όλων των επιπέδων διακυβέρνησης διεθνικό, εθνικό και περιφερειακό. Ο μόνος τρόπος να πετύχουμε τους ε, στόχους αυτούς ε, είναι όχι απλώς να καθορίσουμε κάποιες ε, δράσεις και να, τις, γεμίσουμε τα κουτάκια, αλλά να δούμε πώς στο μέλλον θα έχουμε τις κατάλληλες διαδικασίες για να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Ε, κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς στόχους και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους δικούς συνολικούς στόχους. Ε, οι στόχοι αυτοί έχουν σχέση με όλες τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και συμπεριλαμβάνονται, συμπεριλαμβάνονται δράσεις και σε εθνικό και σε ε, τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν υπάρχει το ζήτημα της επίτευξης των συνολικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ικανότητας του κάθε φορέα που έχει επιφορτιστεί με την υλοποίηση αυτών των στόχων να τους ε, πετύχει. Είναι ελάχιστε οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν που επέλεξαν να μην υποβάλουν νομοδότηση. Αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Αυτό υποχρεώνει εμένα και τους συναδέλφους μου και ως να βρούμε ενδιαφέροντες καινούριου τρόπους να ικανοποιήσουμε όλες τις ε, ανησυχίες. Οι στόχοι αυτοί έχουν επίσης το ρόλο της βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο, στο σύνολό της. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σύντομη, το διατακτικό της είναι, δεν ξεπερνάει τις 800 λέξεις, ε, σε τέτοιου είδου λιτά κείμενα πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος ε, να χάσουμε κάποια ουσιώδη πράγματα. Γι' αυτό το λόγο θα είναι σημαντική η διαδικασία των τροπολογιών. Προκειμένου δηλαδή να δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση σε πράγματα που μπορεί να έχουν ε, μπει στο περιθώριο αυτή τη στιγμή. Τι ήθελα να πετύχω. Η έκθεση θέλει να αποτελέσει το πλαίσιο ενός μελλοντικού οδικού χάρτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο όχι της μόνο της σημερινής μας δράσης αλλά και της μελλοντικής μας. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα με όλους τους ενδιαφερόμενους και τους επηρεαζόμενους γιατί Χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή την πλατφόρμα θα πρέπει να συμμετέχουν όχι μόνο κυβερνήσεις αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Αναφέρομαι σε καθέναν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη Συμφωνία του Παρισιού και την στρατηγική καλύτερης νομοθέτησης. Προσπαθώ να εντοπίσω του τομεί που οι ευρωπαϊκές πολιτικές μας έχουν απομακρύνει από τους στόχου. Για παράδειγμα, παραγωγή βιοκαυσίμων. Τέλος, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι προ αμοιβαιόφελο. Κάποιοι θα χάσουν από τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Ιδιαίτερα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξη και της βιώσιμης βιομηχανίας έχει γίνει της μόδας να ε, επιμένουμε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις που βολεύουν όλους. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα επηρεάσουν με πολύ συγκεκριμένους τρόπους τη βιομηχανία για παράδειγμα. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε να δρούμε με τρόπο μία υφόρο. Κάποιοι κλάδοι θα πρέπει να ε, σταδιακά να καταργηθούν και αυτό θα επηρεάσει πολλούς που εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς και είναι πολύ σημαντικό η μετάβαση να είναι δίκαιη. Πρέπει να τη συζητήσουμε. Άρχισα εγώ ο ίδιος να τροποποιώ την έκθεσή μου. Ορισμένες από αυτές τις τροποποιήσεις, τις τροπολογίες θα τις δείτε και έχουν σχέση με την πλατφόρμα των εμπλεκομένων γιατί μέσω αυτής της πλατφόρμας θα μάθει ένας από τον άλλο. Δεν είναι δυνατόν τα θεσμικά όργανα ο νομοθέτης να ψηφίζει νόμους και αυτοί να εφαρμόζονται τοπικά χωρίς να έχουν να έχει συμβουλευθεί αυτούς που θα, την εφαρμόσουν τους κανόνες. Πολύ συχνά οι δράσεις είναι σε επίπεδο πόλης και πρέπει να αναγνωρίσουμε και, τον, και το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών που έχει εξετάσει το θέμα της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών. Ελπίζω ότι θα δημιουργήσουμε ε, μια πλατφόρμα που τα τρία βασικά, τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητούν το πώς θα εφαρμαλύτερα οι βέλτιστες πρακτικές και εκεί τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας αναφέρουν την εμπειρία τους αλλά και τα βασικά εμπόδια που έχουν συναντήσει. είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε τους στόχους όχι ως επιτροπή μόνο, αλλά και ως κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του το όραμα για την Ευρώπη των επόμενων ετών και δεκαετιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Ποιος Φερία. Να χαιρετήσω τον συνάδελφο κύριο Ντάνς και να τον συγχαρώ. Το προσχέδιο έκθεσης ε, περιγράφει τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχει σχέση με την Ατζέντα 2030 που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική ευκαιρία να εδραιώσει την ηγετική της θέση. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά και προγραμματισμένοι και απαιτητικοί σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Η εποχή μας είναι εποχή αβεβαιοτήτων και πρέπει να βρούμε παρόλα αυτά μόνιμες λύσεις. Ο κόσμος έχει αλλάξει, οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση καθώς επίσης και η κλιματική αλλαγή αποδεικνύουν ότι η οικονομία και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα και δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μία από τις δύο αυτές διαστάσεις χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την άλλη. Το λέει και ο κύριος Ντάνς στην έκθεσή του. Εγώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι, διότι αυτά που προτείνονται είναι πολύ σημαντικά. Να, θα ήθελα να εμβαθύνουμε την πολιτική θεώρηση της έκθεσης. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα δράση πολύ συγκεκριμένο, ε, που θα έχει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στο κέντρο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγκυρωμένα στην Ατζέντα 2030. Οι στόχοι αυτοί καλύπτονται ήδη από δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, μην, ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν είναι επαρκή για να επιτευχθούν οι στόχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Σε γενικέ γραμμέ, η έκθεση αυτή προτείνει και εντοπίζει μέτρα που θα καλύψουν, θα συμπληρώσουν τα κενά των πολιτικών που ακολουθούμε μέχρι τώρα, καθώς επίσης και την κακή εφαρμογή πολλές φορές. Θέλουμε να προωθήσουμε συνεκτικές και σφαιρικές πολιτικές, πολιτικές μακροπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, προτείνει μηχανισμούς συντονισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων και των δράσεων, έναν πίνακα ε, μετρήσιμων δικτών για να αξιολογούμε τους, ε, την πρόοδο στους διάφορους στόχους. Ε, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι οι θεμελιώδεις αρχές της Ατζέντα ε, 2030 θα ενταχθούν Πλήρωση στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω, για παράδειγμα, ενός ρεαλιστικού και συγκεκριμένου προγράμματος δράσης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 22 Φεβρουαρίου 2016 τα επόμενα στάδια για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον επαναλαμβάνει τις αρχές, την αρχή της ε, βιώσιμης ανάπτυξης σε συνδυασμό με την Ατζέντα του 2030. Όμως, δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς η Ατζέντα 2030 θα συγκεκριμενοποιηθεί. Η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία μιας ε, ε, πολυμερούς πλατφόρμας για να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να παρακολουθείται η υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε όλους τους κλάδους, σε επίπεδο κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν αναφέρει τίποτα άλλο για αυτήν την πλατφόρμα. Αυτά θα ήθελα να συμπεριλάβουμε στην έκθεση μέσω τροπολογιών και σε στενή συνεργασία με τον συνάλφο εισηγητή. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εδώ και καιρό στο κέντρο της ευρωπαϊκής δράσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για να προασπίσει τον πλανήτη μας και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κιμπράντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σεπ Ντάνς για την έκθεση που μας έχει υποβάλει. Θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση της Επιτροπής. Συνήθως είμαι θετικός όταν απευθύνομαι στην Επιτροπή. Αλλά πραγματικά έπαθα σοκ διαβάζοντας αυτό αυτή την ανακοίνωση. Είναι εξαιρετικά αδύναμη. Παραδείγματο χάρη είναι ο τίτλος «Επόμενα βήματα για μια εφορία». Πραγματικά εκπλήσωμαι και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάνει την ουσία αυτού του θέματος. Διότι συγκρίνει τους στόχους της χιλιετίας με αυτό. υπάρχει μια τεράστια ουσιώδης διαφορά ότι τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρονται στη μείωση της φτώχειας μιλώντας για την απαραίτητη προϋπόθεση να προχωρήσουμε προς μια αειφορία στην οικονομία. Αυτό που κάνει η Επιτροπή είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή προσπαθεί να δει που αυτοί οι στόχοι έχουν κάποια κοινά με τις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, τα κοινά είναι ελάχιστα. Ε, έχουμε τεράστιε προκλήσεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να καταπολεμήσουμε τη γύρανση του πληθυσμού, να αντιμετωπίσουμε τους πρόσφυγες, το θέμα της Συρία. Μία όμως πάρα πολύ σημαντική πρόκληση είναι να υπάρξει πραγματική μετάβαση προς αηφορία στην οικονομία. Αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα άλλα. Και αυτό το ουσιαστικό σημείο το παρακάμπτει, το χάνει εντελώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πραγματικά αυτό που περιμέναμε ήταν να έρθει ο αρμόδιος Επίτροπος αλλά και ο πρόεδρος Επιτροπής με μία ημερήσια διάταξη που να περιλαμβάνει προτάσεις που να βρίσκονται στην καρδιά όλων των πολιτικών και να οδηγούν προς αυτό το στόχο της αηφορίας. Παραδείγματο χάρη, κοιτώ τη σελίδα 7. Δεν θα υπάρξει αηφορία εάν παραμείνει η ανάπτυξη στα σημερινά επίπεδα. Ναι, το ξέρουμε. Το κοινωνικό μας μοντέλο δεν μπορεί να γίνει αηφόρο και βιώσιμο παρά μόνο αν η οικονομία αποκτήσει βιωσιμότητα και αηφορία. Δεν έχει καμία σχέση με το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Μιλούμε για την αηφορία. Όταν ο Τραμπ λέει America first, εμείς δεν χρειάζεται να απαντήσουμε Europe First. Πρέπει να απαντήσουμε αηφορία κατά πρώτο λόγο, sustainability first. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και η μόνη εγγύησή μας, η μόνη ασφάλειά μας που μπορεί να μας προστατεύσει από εδώ και πέρα. Και τι κάνει η Επιτροπή, τίποτα, απολύτως. Ο Επίτροπος Βέλα κάτι προσπαθεί να κάνει, κάπως κινητοποιείται, αλλά δεν αρκεί. Και πραγματικά είναι εξαιρετικά απογοητευτικά αυτά που μας υποβάλλει εδώ η Επιτροπή. Επιμένω και το υπογραμμίζω με τέτοια ένταση σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε το Brexit. Έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά στην ημερήσια διάταξη. Και η σημαντική ευκαιρία που έχουμε είναι να ανατρέψουμε αυτή την αρνητική ατζέντα επανέρχομαι στο θέμα της ΕΦΣΥ. Θα πρέπει σε όλες τις επενδύσεις, σε όλες τις επενδύσεις παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ΕΦΣΥ, να έχουν σαν προϋπόθεση την αηφορία, την βιωσιμότητα. Δεν είναι δυνατόν εδώ να υπάρχουν επιπλέον δαπάνες και να μην κάνουμε τις σωστές επενδύσεις. Για την ΕΦΣΥ λοιπόν η απάντηση είναι όχι. Το ίδιο και για την κοινή πολιτική. Τραγική κατάσταση. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ βλέπουμε την Επιτροπή υποβάλλει μια γενική στρατηγική για τη βιωσιμότητα που απλώς περιλαμβάνεται στον τίτλο, τίποτα παραπάνω. Κοιτώ λοιπόν την Επιτροπή και ίσως όταν μας υποβάλλει κάτι το ουσιαστικό να μπορέσουμε και εμείς να αρχίσουμε τη δουλειά μας. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε εδώ τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς να έρθει να μας εξηγήσει γιατί πρέπει να χάνουμε την ώρα μας με αυτού του είδους ανακοινώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον προηγούμενο ομιλήτη. Τον Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τη βιωσιμότητα και τις ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη βιωσιμότητα, στην έλλειψη βιώσιμων ε, πηγών ενέργειας, στην γενικότερη πολιτική. Και πραγματικά είναι απογοητευτική αυτή η ανακοίνωση της Επιτροπής, χωρίς όραμα, χωρίς καμία πολιτική απάντηση. Εντοπίζονται κάποια προβλήματα και καμία ε, λύση για να τα ξεπεράσουμε βλέπω την Επιτροπή να ασχολείται με την ε, βιωσιμότητα αγνώντας τα βασικά προβλήματα. Δεν είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή το θέμα της αηφορίας. Θα πρέπει κανονικά να είναι το βασικό ερώτημα. Ναι ή όχι στη βιωσιμότητα, από αυτό εξαρτάται το μέλλον του πλανήτη μας. Για την επόμενη δεκαετία λοιπόν δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να ασχολιόμαστε με αυτό το θέμα. 77% αν θέλετε αυτού από το οποίο εξαρτάται η ζωή μας απειλείται αν δεν υιοθετήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και η διατροφή μας και το περιβάλλον μας και οι πρακτικές για την επιδείνωση, αν θέλετε, της ποιότητας του εδάφους. Μειώνουμε τη βιοπικιλότητα, συρρυκνώνουμε τα είδη, την Φλωρίδα και την Πανίδα. Και πραγματικά εδώ είναι εξαιρετικά επικίνδυνο το να αγνοούμε, παραδείγματο χάρη, την ειδική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που θέτει πάρα πολύ συγκεκριμένους στόχους και που πρεσβεύει μία μεταρρύθμιση και μία αλλαγή και του τρόπου παραγωγής και του τρόπου κατανάλωσης να ενισχυθεί το greening στην κοινή αγροτική πολιτική. Δεν αρκούν όμως όλα αυτά. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπόεβαλε εδώ ένα πάρα πολύ επιφανειακό και αδύναμο κείμενο. Άγνοια για, την, για μένα διακατέχει αυτή την ανακοίνωση και αυτή η τρογική άγνοια θα πρέπει εδώ να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Εκ. Και τώρα συμπαθάτε μου, αλλά θα πρέπει ο υποφαινόμενο να λάβει το λόγο. Τι να κάνω, δεν περίμενα ότι θα αναλάβω την Προεδρία ε, τη στιγμή αυτή. Φυσικά και εγώ θα τηρήσω το χρονικό όριο, οπότε πρώτα πρώτα και εγώ, όπω και άλλοι συνάδελφοι, να πω ότι απογοητεύτηκα ελαφρώ από την Αγίωση τη Επιτροπή, γιατί απέχει πάρα πολύ από αυτό που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε να πετύχουμε τους ελληνικού μας βιώσιμους στόχους και επίση να προχωρήσουμε ευθυγραμμισμένοι με αυτή την πόλη και βέβαια μπράβο στον εισηγητή είναι πολύ ε, καλή η έκθεση και να δούμε επομένω πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ιδίω Εκεί που η έκθεση απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στους ε, στόχους του κλιματολογικού, σχετικό κανονισμό. Αυτούς τους σημερινούς στόχους και τις πολιτικές να προωθήσει που έχουν σχέση με τους στόχους μας αλλά και τις μέσες μας του Παρισιού. Επίσης για την κυκλική οικονομία υπάρχουν ε, κάποιες παραπομπές, ε, αλλά επίσης και για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Μα δεν αρκεί να είμαστε μόνο λόγια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δέσπιση νέων ρυθμίσεων. Επίσης, σε κάποια σημεία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την έκθεση. Αυτό που χρειάζεται πρώτα πρώτα πλευρά τη Επιτροπή να γίνει κάποιο είδου έλεγχο, ανάλυση όλων των πολιτικών τη χρηματοδότηση προ τα κράτη-μέλη σε σχέση με το εάν ευθυγραμμίζονται οι ενέργειες αυτές οι σχετικές με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Τέτοιο έλεγχος πρέπει να γίνει, να δούμε αν η κάθε επιμέρου πολιτική, ο κάθε τομέα μας βοηθά στο να πετύχουμε τους στόχους μας ή όχι. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, αξιολόγηση της πολιτικής για το περιβάλλον αλλά νομίζω ότι οι σχετικές στρατηγικές δεν είναι τόσο αποτελεσματικέ αφήνουν υπερβολικά μεγάλο περιθωρισμό στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται πιο αυστηρό έλεγχος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση να είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά το θέμα τη βιοποικιλότητας. Ξέρουμε ότι πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα. Για τη βιωσιμότητα. Η φυσική μας πόρη, τα οικοσυστήματα κινδυνεύουν. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα να τα προστατεύσουμε, να έχουμε πιο δυναμικές στρατηγικές και καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των ισχυών των μέτρων. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που θα τα συζητήσουμε στις συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις Για το πόσο πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, να περάσουν τα μήνυματα μέσα από την παιδεία. Γιατί σε πολλά σημεία είχαμε πίσω γύρισμα από πλευράς κάποιων κυβερνήσεων, αλλά κυρίως από κοινωνίε σε σχέση με τη βιωσιμότητα, θα πρέπει να επενδύσουμε εκεί πέρα, στην ενημέρωση, στην πειθό του κόσμου, ότι μόνο με βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία μπορούμε να έχουμε κάποια πιθανότητα να έχουμε πετυχημένη οικονομία για την ε, επόμενη μέρα. Η κυρία Εύη, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα πω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Ντάνς. Και εγώ όμως εξίσου θα επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια πρώτη μου σκέψη για τα δεδομένα, τα στοιχεία επί των οποίων βασίζεται η αξιολόγηση πρώτον την υπηρεσία περιβάλλοντος για, για το 16. Αυτό ήταν η αφετηρία μας. Νομίζω ότι το σκηνικό εκεί είναι πάρα πολύ θλιβερό. Και προκύπτει ότι τέσσερις από τους 30 δείκτες δείχνουν επιδείνωση των πραγμάτων για πολλούς τομείς. Α, Φερρυπίν, για τη βιοπικιλότητα, για την προστασία των οικοσυστημάτων, οικοτόπων, για τις μεταφορές. Επίσης, όσον αφορά τα ύδατα επιφανείας, ε, και εδώ υπάρχει έλλειψη στοιχείων. Τα κράτη-μέλη διστροπούν, δεν στέλνουν τα σχετικά στοιχεία. Άρα τι θα γίνει με στόχους του 2020. Δεν θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε, νομίζω δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Έχουμε επίσης 7 άλλους τομείς. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση διαχρονική. Αλλά υπάρχει δυσκολία επίτευξη των στόχων του 2020 και μιλώ για κάποια οικοσυστήματα για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, για τα οξύδια αζόντου που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, την ηχορύπανση, αλλά επίσης και την κατανάλωση ε, ψαριού και κρέατος. Άρα μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε τάξει. Επομένως από τους 30 στόχους Έχουμε εννέα που είπαμε ότι έχουμε κάποια πρόδαστα στα κατά τα λοιπά. Είπαμε θλιβερό το σκηνικό θα πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς η κοινοτική δράση θα πρέπει να γνωρίσει μια νέα δυναμική. Ε, επίσης, να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι ισχύει για τους δείκτες, γιατί πώς μας βοηθάνε για την αξιολόγηση. Συχνά έχουμε κάποιους δείκτες που δεν είναι τόσο ακριβείς. Να, ένα δεικτικό παράδειγμα. Για την ποιότητα της ατμόσφαιρας της πόλης, πολλές φορές έχουμε αυτό το 2,5% αλλά πολλές φορές έχουμε υποτίμηση των ε, άλλων εκθέσεων και επίσης της σημασίας των φίλτρων που μολύνουν με κάποια μικροστοιχεία που εκπέμπουν και άλλους τρόπους μόλυνσης. Όλα αυτά θα έπρεπε να αποτελούν ξεκάθαρους δείκτες στα επίσημα στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ETS, του σύστημα εμπορίας των εκπομπών για πολιτική για το κλίμα. Ήρθε η ώρα τώρα να κάτσουμε και έντιμα και σοβαρά να κάνουμε μια κριτική ανάλυση του τι έχει γίνει. Δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να προσπαθήσουν οι κλάδοι να επενδύσουν εκεί που χρειάζεται, που είναι οι πιο βρώμικοι στους υπηρετηριότητες. Οπότε και πάρα πολλές από τις χρηματοδοτήσεις που διαθέτει η Ένωση πάνε σε κάποια φαρονικά έργα που και άχρηστα είναι και μολύνουν. Και σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα. Ε, δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε, δεν μας πάνε σωστή κατεύθυνση. Η κυρία Ντορνανό είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ στον εισηγητή για την έκθεσή του. Αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολείται με πολλά διαφορετικά θέματα, την οικονομία, τη μετάβαση στην πολιτική της ενέργειας, την ανάπτυξη, όλα αυτά αναμειγμένα χωρίς να προτείνει συγκεκριμένα ότι πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο όσον αφορά τη λειτουργία μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε της σημερινής ε, κατάστασης, την ενταδικοποίηση των ροών εμπορικών και ανθρωπίνων, η αύξηση των ε, αποβλήτων, κυρίως τα πλαστικά, που μολύνουν συγκεκριμένα τους ωκεανούς και τις θάλασσές μας. Η προστασία της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε σήμερα ότι για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για τη νεολική ενέργεια η ευρωπαϊκή οικονομία, η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει εντελώς καταστραφεί από το dumping από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα από τη Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να υπάρξει δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτά είναι κάποιες από τις σκέψεις που θα ήθελα να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική μας συζήτηση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. <coughs> Μετά τους Κιώδης θέλουν και άλλοι βουλευτές να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Νομίζω ότι αρκετή κριτική ακούστηκε μέχρι τώρα για την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ε, πολιτική της αηφορίας. Μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα άκουσα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή, γιατί όλοι εμείς Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε έτσι ώστε να κάνουμε στο ένα βήμα προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Είμαι εισηγήτρια για την Επιτροπή Γεωργίας και διαπίστωσα διαβάζοντα την έκθεσή σας ότι η συγκεκριμένη γεωργία που είναι αρμοδιότητά μου, αλλά συγκεκριμένα και το θέμα των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απασχολεί καθόλου την έκθεση αυτή. Βεβαίως και είμαστε εδώ υπεύθυνοι για χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στον τομέα της γεωργίας και της δεσοκομείας στην ε, Γερμανία. Το 1 τρίτο των ε, εκτάσεων της γης που είναι αφιερωμένες στην καλλιέργεια, στη γεωργία ανήκουν σε κάποιες από τις πολιτικές, από τα προγράμματα προστασίας, περιβαλλοντολογικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η δική μας δράση και την ίδια ώρα πρέπει να προστατεύσουμε όλους όσους εργάζονται στον τομέα αυτό, όλους όσους εργάζονται στον τομέα της βιωσιμότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και την ίδια ώρα θέλουν να κερδίσουν να ζήσουν συγγνώμη, από τη δραστηριότητα αυτή. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βλέπουμε την οικονομία αποκομμένη από την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες και ήθελα να ενημερώσω τον συγκητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντάλη. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πρέπει να επιβεβαιώσουμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης όπως αναφέρονται στην Ατζέντα 2030 των ΗΕ. Ο εισηγητής, ο κύριος Ντάντς ε, έχει δύσκολο έργο. Παρ' όλα αυτά, το κείμενο που έχει προετοιμάσει ως προσχέδιο είναι πολύ καλό και νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε ως βάση για να αναπτύξουμε τις ιδέες μας. Εμείς ως πολιτική ομάδα πιστεύουμε ότι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης είναι πολύ επίγον να ε, τύχει επεξεργασίας και να εξειδικευτεί σε κάθε τομέα της δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Αυτά προκειμένου να σταθούμε στο ύψος των φιλοδοξιών της Ατζέντα 2030. Πρέπει να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους χρειάζεται περισσότερη δράση και το συντομότερο δυνατό να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται. Θα πρέπει επίσης ε, να λάβουμε υπόψη μας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσει το μεταναστευτικό. Γιατί αυτό αποδεικνύει ότι η έλλειψη βιώσιμης ανάπτυξης σε άλλα μέρη του κόσμου μας δημιουργεί προκλήσεις. Το θέμα επίσης συνδέεται με διαφορές στις οικονομίες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις διαφορές. Χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση, συνοχή για την πολιτική ε, βιώσιμη ανάπτυξη ανάπτυξης σε άλλου τομεί, όπως ο τομέα, το μέσο των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας. Οι αποφάσεις μας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν τα κείμενα τα οποία εγκρίνουμε εμείς ως νομοθετήματα. Αυτά τα κείμενα τα θα επηρεάσουν και τη ζωή των, τη δική μας αλλά και των παιδιών μας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορούμε να στρέψουμε το βρέμα προς τα πίσω και να είμαστε περήφανοι για τις αποφάσεις που είχαμε πάρει. Ελπίζω ο εισηγητής με τους εισηγητές να καταφέρουν να μας προτείνουν μια έκθεση που θα είναι ισχυρή και θα ε, αντιμετωπίζει τα παλιότερα προβλήματα επικοινωνίας που είχαμε. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν τώρα έχει το λόγο, κύριε Σμάκελ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ε, καταγράφω τις ε, κριτικές σας. Για μας η έκθεση αυτή καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα σχετικά ζητήματα. Και είναι και πάρα πολλά, διότι το είπε και ο εισηγητής και για μας ήταν πάρα πολλά ε, είναι πολύ σημαντικό και εμείς στην ανακοίνωσή μας και ο εισηγητής να υπογραμμίζουμε το, την ποικιλία των ζητημάτων τα οποία καλύπτονται, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καθιστούμε σαφές ότι οι πολιτικές για το περιβάλλον μας μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τη βιωσιμότητα. Όμως, θα πρέπει να δούμε και τη βιωσιμότητα σε κοινωνικό, για παράδειγμα, επίπεδο, ε, σε επίπεδο των δύο φύλων κλπ. Η έκθεση αναφέρεται στην ενεργειακή πολιτική, στην κυκλική οικονομία και στην ανακοίνωσή μας είπαμε ότι το αναφέρουμε θέλουμε να διατηρήσουμε ηγετική θέση για όλα αυτά τα θέματα στο μέλλον. Τώρα, οι συνάδελφοι στήριξαν τις πολιτικές οι οποίες προτείνουμε. Κυρίως εξυγχρονισμό και συνέργειες. Συνεργατικές δράσεις στον περιβαλλοντικό τομέα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, να εργαστούμε πλάι-πλάι και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε για την καλύτερη νομοθέτηση όπως για παράδειγμα το Project Team, την ε, ομάδα, διυπηρεσιακή ομάδα της ε, Κομισιόν για κάθε συγκεκριμένο project τρέχει. Τώρα, όλα αυτά έχουν σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη διαδικασία της Λευκής Βίβλου που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν. Δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή να σας το αναπτύξω. Έχουμε όμως πολλές σκέψεις, πολλές ιδέες και θα δούμε κάθε μία από αυτές χωριστά. Τώρα, να σχολιάσω μερικές από τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις που κάνατε. Πρώτον, συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που είπε ο και άλλοι ότι οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό τρόπο σκέψη. Το λέμε και εμεί στην ανακοίνωσή μα. Όλοι μαζί θα πρέπει να συνεργαστούμε σε ένα πιο, με ένα πιο επικοδομητικό τρόπο, με ένα καινούριο τρόπο. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη μια πλατφόρμα όλων των μερών και των κρατών μελών για να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και να πάρουμε τι συμβουλές τους. Πολλοί από εσά μιλήσατε για τη σημασία των μετρήσεων. Κρίσιμο σημείο αυτό γιατί έχουμε να δώσουμε λογαριασμό στα Ηνωμένα Έθνη και ως κράτη-μέλη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τους τελευταίους μήνες ε, αναπτύσσουμε δείκτες τους οποίους θα συμπεριλάβουμε στην ε, έκθεση πρόοδου του 2017. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στην ανάγκη προγράμματος δράσης. Στην ανακοίνωσή μας επιλέξαμε να μην ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, γιατί ένα πρόγραμμα εργασία για τα επόμενα 15 χρόνια και για όλους αυτού τους τομεί θα ήταν αδύνατο να γίνει. Όμως θα έχουμε ετήσια προγράμματα δράση τα οποία θα αποδεικνύουν ότι παίρνουμε στα σοβαρά την βιωσιμότητα. Τώρα, τι είπε ο κ. Γκερμπράντι που ήταν πολύ ομός στις κριτικές του, να τα σχολιάσω λίγο. Λέτε ότι δεν έχουμε μιλήσει για την οικονομική μετάβαση. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει. Στο τέλος της ανακοίνωσης λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπει σε καινούργια τροχιά στην παγκόσμια οικονομία. Και αυτή πια είναι η κυκλική οικονομία. Έτσι κι αλλιώ η ανακοίνωση προβλέπει ετήσιο πρόγραμμα εργασία για το οποίο θα υποβάλουμε έκθεση ε, ε, τακτικά. Η κυκλική οικονομία έχει άμεση σχέση με 8 από τους στόχους. Ε, και μόνο 12 ε, στόχοι χρειάζονται καλύτερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, βιοπικιλότητα. Ξέρω ότι έγινε ένα ε, fitness check και στην ανακοίνωση λέμε ότι πρέπει να αναλυθούμε να η δράση. Εκεί και στο πλαίσιο της αρχής των παγκόσμιων συνόρων πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε πηγόντως. Τώρα για τόσο είπε η Ντάλη στο τέλος. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις είναι πράγματι η μετανάστευση. Και η ανακοίνωση εξετάζει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της, αλλά συνοδεύεται και από ένα δεύτερο έγγραφο, το, την Ευρωπαϊκή Συνένεση, ε, η, ο, κάτι το οποίο δείχνει Πώ πρέπει να δούμε και την εσωτερική μα πολιτική και την εξωτερική μα πολιτική, όπω λέμε στην ανακοίνωση. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα ολοκληρώνουμε την συζήτηση. Απευθυνόμενοι και πάλι για δευτερολογία στον κύριο Ντάν. σα. ευχαριστώ όλου για όσα είπατε. Γιατί είπατε ότι είναι πολλά τα στραβά με την ανακοίνωση και συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέλφους οι οποίοι τόνισαν ποια είναι τα δυνατά σημεία. Αλλά μπορεί κανείς να κινηθεί κατά δύο τρόπους. Ίσως καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου διατυπώνουμε ότι υπάρχει τόση έλλειψη φιλοδοξίας που η μόνη επιλογή είναι να ακολουθήσουμε άλλη μεθοδολογία και να προτείνουμε κάτι όλος διαφορετικό. Όμως τώρα μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί αν ανταποκριθούμε στην κατάσταση. Και ξέρουμε όλοι το μέγεθο των προβλημάτων και τη πρόκληση και ξέρουμε τι γίνεται με το, τη μεγάλη φαλοκρηπίδα, το μεγάλο ύφαλο, τον barrier reef. Τον κορελογενή ύφαλο τέλο πάντων. Και αν όλα αυτά καταστραφούν, τι θα πούμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας, ότι σταυρώσαμε τα χέρια ενώπιον της καταστροφής, ε όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα προδίδαμε όχι μόνο τις μέλους της γενιάς, αλλά και τους εαυτούς μας. Και αυτό που κανείς μπορεί να εντοπίσει αυτά που λέει η Κομισιόν είναι ότι υπάρχει κάποια διαμάχη και εκεί όσον αφορά το πόσο φιλόδοξη θα είναι η πρόταση. Και έτσι το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι όχι μόνο θα υπάρχει μια εξορρόπηση των επιμέρους πραγμάτων, αλλά θα είναι κομισιόν φιλόδοξη, θα έχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται, ούτω ώστε να μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει η κομισιόν. Ε, καλά, δεν, δεν πρέπει κανεί να κατακυλάει και να πει ότι «Α, καλά, ας κάνουμε ό,τι, ό,τι γίνεται». Όχι, ας κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Να δούμε πώς θα γίνει mainstreaming πώς θα εντάξουμε στις πολιτικές τους βιώσιμους στόχους. Αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια. Είναι κάτι που εν υπάρχει θα κάνει η, Επίτροπη. Θα πρέπει και με το ζόρι να γίνει αυτού του είδους η ένταξη. Να μην πάμε περιπτωσιολογικά πρόγραμμα δράσης, ε, έχουμε μετά τους πόρους, μετά έχουμε δύο ποικιλότητα και γεωργία, ε, κατόπιν έχουμε το μεταναστευτικό, διαφορές κρατών μελών. Αυτά είναι γνωστά ότι υπάρχουν, θα πρέπει όλα αυτά να τα συγκεράσουμε, θα πρέπει αυτά ως προτεραιότητες να αντανακλώνται στην έκθεση. Να μην έχουμε μια παραδοσιακή προσέγγιση και ο τελικά ο καθένας να θέλει να περάσει τις θεσούλες του και να πάρει κάποιους πόντους. Βεβαίω και εδώ αιτία είναι και αυτή η ματιός που νιώθει κανεί. Ε, αυτή η απογοήτευση για αυτή την ανακοίνωση της Κομισιόν ευθύ εξ αρχής. Από την άλλη μεριά όμως τα θεσμικά όργανα είναι φιλόδοξα. Ε, αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου, εν και γενικότερα. Εμείς πρέπει είμαστε συνεφόροι της φιλοδοξίας. Αυτό να κάνουμε σε την έκθεση. Ας την κάνουμε φιλόδοξη. Και ας συμπαρασύρουμε και άλλους. Ελπίζω αυτή να είναι τελικά η προσέγγιση. Εγώ αυτό πάντως πασχίζω να πω. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε εισηγητά, ευχαριστώ και όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Να σας πω τώρα πώς έχει το χρονοδιάγραμμα. 25 Τετάρτου στις 11 η ώρα. Είναι η προθεσμία για τροπολογίες. Και θα δούμε μετά. 21-22 Ιουνίου να πάμε. Οπότε κλευρώσαμε το σημείο υπαριθμό 7 και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι η αιτήσια συνάντηση για τα απόψεων με τον καθηγητή Hans Brownings, που είναι ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Καθίστε, καθίστε, λέει η Πρόεδρος. So, thank you very much for... Και σας ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνάντησή μας για την ανταλλαγή απόψεων. Θα ζητήσουμε το πρόγραμμα εργασία για το 2017. Ευθύ αμέσω. Σα δίνω το λόγο για να κάνετε την εισαγωγή σα. Και ελπίζω συνάδελφοι θα σκαρφιστούν ερωτήσει και θα ακολουθήσει η συζήτηση από αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ λέει ο κ. Μπράνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτέ, είναι μια αξιόλογη ευκαιρία αυτό κάθε χρόνο να δώσουμε άποψη όσον αφορά το έργο μα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Βέβαια δεν είναι αυτή η μόνη μα συνεργασία, η ημών και ημών. Γιατί ήδη σα ανέφερα ότι επανειλημμένα έχουμε έρθει σε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ εδώ, στην ΙΜΙΣ, στην Τρασπορ, στην Επιτροπή Ενέργειας, και ενημερώνουμε τι, τι, δουλειά κάνουμε σε σχέση με τις πολιτικές που ασκούνται. Επίσης, κάποια στιγμή συναντηθήκαμε στην ετήσια επίσκεψη που κάνατε στην υπηρεσία μας, στην Κοπενχάγη. Ήταν παραγωγική αυτή η επίσκεψη, ήρθαν οι πολλοί βουλευτές, συναντήσαμε τη νέα πρόεδρο, αλλά και την γραμματεία τώρα πρόσφατα και είπαμε ότι θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε συγκεκριτές και σκιώδες συγκεκριτές, εάν το θέλουν βέβαια. Βέβαια, ο μπούσουλας μας είναι το πολιτές πρόγραμμα. Θα πρέπει να δούμε πώς η εφαρμογή των πολιτικών θα βασίζεται στη γνώση, αλλά και σε κάποιο είδους μετάβαση, μετασχηματισμό μακροπρόθεσμο, γιατί έχουμε το, το κεκτημένο και τελικά να έχει κάποιο νόημα. Και έτσι να μπορούμε να βοηθήσουμε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά αλλά κυρίω να μπορούμε να βοηθήσουμε του συνεργαζόμενου, αλλά κυρίω κυρίως τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα και τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον που είναι η προσταμένη μα αρχή κατά κάποιο τρόπο. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και προ πιο ολοκληρωμένο θεματολόγιο ε, εν ώψη του 2030 και του 2050. Ε, και έτσι προβλέπονται τι αλλαγέ θα γίνουν όσον αφορά τα στήματα παραγωγή και κατανάλωση. Αυτά τα θεματολόγια έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχω να σα πω ότι όταν εγώ ανέλαβα το 2013, και φτιάξαμε αυτό το πολιτικό πρόγραμμα. Δεν υπήρχε τότε κανένα, κανένα πακέτο ε, κυκλική οικονομία, δεν υπήρχε καμία σημαίνει των Παρισίων, δεν υπήρχαν στόχοι διόρθμιση ανάπτυξη. Οπότε και έτσι ετησίω προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε επί τη βάση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίση δεν πρέπει να ξεχνούμε το ότι πρέπει να δίνουμε προσοχή κυρίω στο τι γίνεται με τα κράτη-μέλη. Γιατί συνεργάζονται και βοηθούμε και του 28 ε, που είναι μέλη στην υπηρεσία μας τους ε, βοηθούμε. Βοηθούμε να αναπτύξουν δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο με τα δικά τους θεματολόγια. Τώρα, για να δούμε σύντομα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στρατηγικούς τομείς του έργου μας. Πρώτα-πρώτα, η πολιτική ενημέρωση που έχει σχέση βέβαια και με την υλοποίηση του κεκτημένου. Πρώτα-πρώτα, ε, ατμοσφαιρική ρήπανση και όσον αφορά ε, την ετήσια έκταση για την ποιότητα του, της ατμόσφαιρας, όπως επίσης και τις εθνικές οροφές των εκπομπών. Και εδώ ότι θέλουμε να υπάρχει μια ποιοτική συζήτηση σε κρατή μέλη. Αυτό είναι ψηλά στο θεματολόγιο και οπότε ευχαρίστω και εμείς να βοηθούμε με κάποιο είδους θεμελιώδη δεδομένα και με την απαιτουμένη ανάλυση και σας τονίζω προκειμένου ότι όλο ένα και περισσότερο συσχετίζουμε το έργο μας με τα θέματα υγείας, με τα θέματα οδήγησης, μεταφορών, ε, ποιότητα ατμόσφαιρας. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία για τι βιομηχανικέ εκπομπέ, όσον αφορά τι εκπομπέ ε, ρηπαντών και το σχετικό μητρό, είπαμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτά στι πολιτικέ, γιατί θεωρούμε ότι θα βγούμε κερδισμένοι σε επίπεδο των μελών και σε επίπεδο ένωση. Τώρα όσον αφορά το πλαίσιο της ενεργειακής ένωσης, θα βοηθήσουμε την διακυβέρνηση στους τέσσερις τους πέντε πυλώνες για τις εκπομπές ε, θερμοκηπίου, ανιώσιμες πηγές ενέργειας, ε, πλασματική χρήση ενέργειας και όσον αφορά το πακέτο ενέργειας και για το 2020 έχουμε τις ε, αναφορές εκθέσεις κατών μελών και κοιτάμε αν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους 2020, κατόπιν έχουμε την πλατφόρμα ADAPT, κλίμα ADAPT. Συνεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτή την ε, προσαρμογή και θα πρέπει να πούμε ότι λόγω του ότι ήδη ζούμε τις αλλαγές στο κλίμα και έχουμε αυτή την τετραετή έκθεση για τα ευάλωτα, για τις επιπτώσεις στην Ευρώπη, το θέμα της προσαρμογής μετά συνέχεια των Παρισίων είναι ένα μέτωπο το οποίο το προσέχουμε όλο ένα και περισσότερο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σχετικά όργανα και κράτη-μέλη για αυτή την πλατφόρμα. Επίσης, ασχολούμαι με ένα σημαντικό νομοθέτημα, ασχολούμαι εντατικά φέτος. Γιατί έχουμε την έκθεση του 2017 ε, ε, για το νερό. όσον αφορά την μόνιση του νερού, όσον αφορά την τους οικοσυστημικούς ε, στόχους που ε, ακόμα επιδέχονται καλύτερη επιδόσεις. Επίσης το σύστημα πληροφόρησης για την Ευρώπη, αυτό αφορά τους πάντες, εμπλέκονται και οι πολίτες και εδώ πέρα είναι το θέμα αυτής της στρατηγικής μετά για τη θάλασσα. Υπάρχει σχετική οδηγία. Οπότε χρειάζεται και περισσότερο να αναγνωριστεί ο ρόλος των θαλασσιών οικοσυστημάτων, αλλά και το πόσο κομβική σημασία έχουν για το, το κρατός, κάθε κρατός μέλος, για την αλλαγή του κλίματος. Οπότε ήδη ετοιμαζόμαστε για το 2019 που θα έχουμε την σχετική έκθεση για το πώ έχουν τα πράγματα για την θάλασσα. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική τη βιοποικιλότητας. Είμαι σύντομος, διότι γνωρίζετε την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα για τα οικοσυστήματα και για τις ε, οδηγίες που αφορούν τα οικοσυστήματα, τη βιοπικιλότητα. Στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση όλους τους οργανισμούς αυτούς που εργάζονται και δραστηριοποιούνται ναι. στον τομέα αυτό. Τέλος, ο έλεγχος όσον αφορά την ε, οδηγία που αφορά κάθε περίπτωση την μείωση του βάρους εργασίας, του όγκου εργασίας και βεβαίως το γεγονός ότι θα πρέπει κάθε φορά να συμμορφωνόμαστε με τα προαπαιτούμενα της ε, νομοθεσίας. Θα ήθελα να μιλήσω και για την κυκλική οικονομία, για την αποτελεσματικότητα των ε, φυσικών πόρων. Εδώ κάνουμε Αποκινούμε άλλους επιστημονικούς οργανισμούς ε, στα κράτη-μέλη, κοινέ μελέτες με τη Eurostat και με τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον κυρίως. Θεωρούμε ότι εδώ πρέπει να καλύψουμε ένα σημαντικό χάσμα που συνεχίζει να υπάρχει όσον αφορά τη γνώση, τα στοιχεία που διαθέτουμε για την κυκλική οικονομία. Ξεκινήσαμε πέρσι και θεωρούμε ότι το χάσμα αυτό θα καλυφθεί και όσον αφορά τη γνώση που έχουμε, αλλά και τους τομείς τους οποίους ακόμα μας λείπουν πολλά στοιχεία. Το θέμα της μετάβασης που αφορά την βιωσιμότητα από το 2013 μέχρι το 7ο πρόγραμμα δράσης ε, εργαζόμαστε και για όλες ε, τις ε, πολιτικές, τη στρατηγική που αφορά τα συστήματα ενέργειας, την ατζέντα για μια μετάβαση σε σύστημα κινητικότητας που να έχει αηφορία, θέματα που αφορούν τις μεταφορές, τα είδη διατροφής, τη γεωργία και ενίσχυση των δυνατοτήτων μας που αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική και τη μεταρρύθμισή της, την ανάλυση που θα ακολουθήσει, τη λεγόμενη Urban Agenda, την ατζέντα του Άμστερνταμ που αφορά τη βιωσιμότητα και την αηφορία στην Ευρώπη. Κάποιος ε, είπε προηγουμένως ότι βεβαίως βασιζόμαστε στους δείκτες, μελέτη βάση δείκτων, και μια οικονομία που να βασίζεται σε περιορισμένες εκπομπές ε, σε άνθρακα, καθώς και την αποτίμηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων για την δημόσια υγεία. Εχθές ξεκίνησε η νέα μελέτη, την έχουμε ξεκινήσει η προεκτική μελέτη μέχρι το 2020, η υλοποίηση του κεκτημένου με τις 17 προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη μετάβαση, ιδιαίτερα σε συστήματα χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και την ενεργειακή μετάβαση. Η λεγόμενη Human Biomonitoring Initiative, η πρωτοβουλία HPM4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξεχνεί στη Γερμανία και που θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε νέες ε, προκλήσεις σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας. Πρόεδρε, συνεργαζόμαστε επίσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης για να βελτιώσουμε την γνώση μας. Ε, επίσης στο ε, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρητηρίου ε, για, την, για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το AONET. Τα δύο επόμενα χρόνια θα ασχοληθούμε πολύ με το ReportNet που είναι η ραχοκοκαλιά από τεχνολογικής πλευράς στην αναφορά περιβαλλοντικών, στις αναφορές περιβαλλοντικών στοιχείων Εκεί καινοτομούμε και σε θέματα ασφάλειας του ίντερνετ. Επίσης ε, συνεισφέρουμε και στο θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω πιο πολύ από την πλευρά του αξιολόγησης ενώ γύρω στα πλευρά των αριθμητικών στοιχείων και βέβαια έχουμε και την χερσία πτυχή του Κοπέρνικος ε, ε, και της ε, ποιότητας του αέρα. Στην ε, νότια γειτονία έχουμε την στρατηγική για τη Μεσόγειο και συνεργαζόμαστε με τις χώρες του Νότου, με τις χώρες της Ανατολής συνεργαζόμαστε κυρίως σε θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης συνεργαζόμαστε να με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τέλος, Στη τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια αξιολόγηση ε, με τους κανόνες του fitness check κάτι που σημαίνει ότι θα ε, αξιολογηθούμε με τα πέντε κριτήρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση του κανονισμού μας και της αποστολής μας ε, και βέβαια μπορεί να έχει και επιπτώσεις στο προσωπικό μας, ε, μισθούς κλπ. Σε ό,τι αφορά τους, ε, τα πρόσθετα καθήκοντά μας, ανεφέρθηκα σε σχέση με ορισμένα από αυτά για, από το 2013 και μετά. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες ώστε να έχουμε τους απαραίτητους πόρους και τέλος αρνητικές προτεραιότητες. Το 2013 είχαμε προβλέψει 5% μείωση στο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ε, μείωση κατά 10% του προσωπικού ήδη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται, χρειάστηκε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητε μας. Ε, όχι με χαρά. Ε, Ήμασταν υποχρεωμένοι όμως να κάνουμε αυτού του περιορισμού στι δραστηριότητέ μα, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε καλή ποιότητα στη δουλειά μας. Μεταξύ αυτών ε, των περιορισμών έχουμε περικόψει τη διεθνή μας συνεργασία, δεύτερον, περιφερειακή συνεργασία, σε ό,τι αφορά περιφερειακές θάλασσες και συμβάσει των ωραίων, Επίσης, περιορισμός της δραστηριότητας μας για τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς επίσης και, τον, και την παρουσία μας στις Βρυξέλλες. Σχεδόν κάθε μέρα κάποιος υπαλληλός μας δουλεύει εδώ στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς πια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην ίδια ένταση και στο ίδιο βεληνικές. Επίσης περικοπές θα κάνουμε και αλλού Ειλικρινά σας λέω, αν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα, δεν θέλω να επενδύσω κάπου. Αφόσον έχουμε λιγότερους πόρους, θα κάνουμε και λιγότερα πράγματα, αλλά με την ίδια ποιότητα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αν γίνουν και άλλες περικοπές στον προϋπολογισμό μας, θα πρέπει να το συζητήσουμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο και με εσάς. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ σαφή όλα αυτά, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στο σημείο επαφή με την υπηρεσία που είναι ο κ. Γερμπράντη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Πάντα χαιρόμαστε να σας βλέπουμε και αξίζεται πραγματικά την παρουσία περισσότερων συναδέλφων. Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσω περαιτέρω. Η η υπηρεσία σας είναι από τις πιο σημαντικές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο από αυτά που είπατε. Ότι περισσότερες περικοπές θα επηρεάσουν την ποιότητα του έργου σας. Εγώ θα το πω ανάποδα. Αν πιστεύουμε ότι το έργο της υπηρεσίας περιβάλλοντος είναι σημαντικό. Θα πρέπει να αποφύγουμε περικοπές και να αυξήσουμε μάλιστα τον προπολογισμό σας. Γιατί η υπηρεσία σας έχει αυτή τη στιγμή λιγότερο προσωπικό από ό,τι πριν από 10 χρόνια είναι δύσκολο κανείς να το εξηγήσει. Ενώ κράτη-μέλη και κομισιόν έχουν αναλάβει περισσότερα, μάλλον έχουν αναθέσει περισσότερα καθήκοντα στην υπηρεσία περιβάλλοντος. Αν δούμε μάλιστα και τις ε, διεθνείς εξελίξεις, αποδεικνύεται ότι ο ρόλος της υπηρεσίας περιβάλλοντος έχει αυξηθεί. Πώς λοιπόν μπορεί η υπηρεσία να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις απαιτήσεις των καιρών. Οπότε η ερώτηση μου είναι εξή. Υποχρεωθήκατε να μειώσετε τις εργασίες σας σε σχέση με την διεθνή συνεργασία. Η, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, μπλοκάρισαν ε, οποιαδήποτε αφορά στη Συμφωνία του Παρισιού στο, στα συμπεράσματα της G7, του G7. Ταυτόχρονα η υπηρεσία, ε, η υπηρεσία περιβάλλοντος των Πολιτείων είδε τον προπολογισμό της να μειώνεται κατά 30-40%. Η συνεισφορά των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη επίσης θα μειωθεί. Πολύ. Οπότε η ερώτησή μου είναι εξής μείωση της διεθνούς συνεργασίας από μέρους σας. Και ταυτόχρονα όλες αυτές οι αρνητικές εξελίξεις από πλευράς των ΗΠΑ τι σημαίνουν. Η, από ό,τι φαίνεται σημαίνει ότι και οι δύο βασικοί συνεισφέροντες ε, στα περιβαλλοντικά θέματα παγκοσμίω, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνουν τη δράση τους. Επίσης αναφέρατε την διαδικασία αξιολόγησης. Είναι εξαιρετικά σημαντική. Γιατί το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν για την υπηρεσία σας. Τέλος, μια πρόταση. Η κυκλική οικονομία γίνεται όλο και πιο σημαντική έχουμε την κατάσταση του περιβάλλοντος, την κατάσταση της φύσης. Δεν θα πρέπει να υποβάλλεται και μια έκθεση για την κατάσταση της κυκλικής οικονομίας, μήπως. Πάλι βέβαια θα σας αναθέτουμε περισσότερα καθήκοντα, αλλά από πλευράς περιεχομένου θα ήταν πολύ σημαντικό. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε το ζήτημα. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα. Μόνο και δεν τα λέγει ζητήσει λόγο. Τι τον δίνω αμέσω. Κάποιο άλλος, α, ο κύριο Σεκ, α, ο κύριο Γιάβορ, α, ωραία, σηκώστε το χέρι σα και η Γερμανιάνο πρόκειται να καταγράψει το έτοιμά σα. Ντάλι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Μπράουνι που ήρθατε και μας κάνατε αυτή την εισήγηση. Δεν μου άρεσε αυτό το τελευταίο που αναφέρατε και που μας είπατε το πόσο στριμωγμένοι είσαστε οικονομικά. Και εγώ στεγόμαι σε αυτό γιατί για μένα σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα. Θα πρέπει να καταλάβουν τη σχέση ευημερία του κόσμου και περιβάλλοντος. Δηλαδή τη σχέση περιβάλλοντος αλλά και την κατάσταση της δημοσίας υγείας του πώς είναι σήμερα η κατάσταση και πού μπορούμε να φτάσουμε καλύτερα. Και αυτό το σκέφτομαι ακριβώς ακούγοντας αυτά τα οποία εσείς μας είπατε στο τέλος. Πάντως εγώ θέλω κάτι άλλο να αναδείξω, το οποίο έχει σχέση με το περιβάλλον και την δημόσια υγεία των συμπολιτών μας. Και εσείς το αναφέρατε στο σημείο που μας είπατε για την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας και τις εθνικές οροφές εκπομπών. Σχεδόν κάθε μέρα βγαίνουν στο φως μελέτες που συνδέουν ε, την μόλυνση των πόλεων με τις ασθένειες, με τους κινδύνους για την υγεία κατά των πολιτών και του που συνδέονται με τις οδικές μεταφορές και έχουμε μία μελέτη του 16 της ε, υπηρεσίας περιβάλλοντος. Τότε τη δημοσίευατε και είπατε ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι υψηλής ποιότητας και επομένως εγκυμονούνται κίνδυνοι, κίνδυνοι για την Ευρώπη. Στην έκθεσή σας επίσης είπατε ότι οι μειώσεις των εκπομπών τα πάνε καλύτερα. Έχει βελτιωθεί η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε ακόμα τη βλάβη στην υγεία και στο περιβάλλον. Μια που μας μιλάτε για την, το κόψιμο του άνθρακα από τις οδικές μεταφορές, βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωράει προς μια φάση όπου θα έχουμε την επανάσταση του ηλεκτρονικού οχήματος στα κράτη-μέλη. Α, στην Ορβηγία, Φερρυπίν. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς τα ίδια. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει σε, σε, επίπεδη πολυεπίπεδη αντιμετώπιση τη κυβέρνηση. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποια διαβήματα και να υπάρχει τελικά θετική ε, επίδοση σε αυτά. Ή πρόεδρο. Ευχαριστούμε κύριε Γιάβορ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε Χάνης που ήρθες να μας επισκεφτεί σήμερα. Όπως ε, προείπαμε, πάντοτε σε βλέπουμε με ευχαρίστηση να ανταλλάσσουμε απόψεις και συμφωνώ ότι είναι ανησυχητικά αυτά τα οποία είπες ότι μάλλον θα υπάρξουν περικοπές στο κονδύλιο για την υπηρεσία σας. Οπότε δεν ξέρω, τώρα ίσως δεν είναι τόσο εύστοχο να πω αυτό που θέλω να πω. Ήθελα να πω για αύξηση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Γιατί τα είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση που νομίζω ήταν εδώ και τα ακούσατε. Τώρα που συζητούσαμε το θέμα των στρατηγικών στόχων ανάπτυξη. Νομίζω ότι πέραν όλων των άλλων έχουμε τώρα δύο σημαντικά θέματα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Πρώτα πρώτα την εφαρμογή των ισχυών των κανονισμών, γιατί επανειλημμένα είδαμε ότι πολλές φορές έχουμε πάρα πολύ άρτιους κανονισμούς, αλλά όταν έρχεται η ώρα της μεταφοράς ιστορικού δίκαιου, όταν έρχεται η ώρα της όσον αφορά την εφαρμογή από τις αρχές, ε, τότε αλλού καταλήγουμε. Αλλού από ότι τι σκεφτήκαμε όταν φτιάξαμε τον κανονισμό. Αυτό και, και για την αξιολόγηση της πολιτικής για το περιβάλλον. έχετε συμμετάσχει, αλλά εσείς βλέπετε να έχει η υπηρεσία σας κάποια περιθώρια να συμμετάσχει πιο ενεργά, πιο δυναμικά στους ελέγχους, στο τι κάνει η Ένωση, σε ό,τι κάνει η Κομισιόν που είναι ο φύλακας των συνθήκων. Να μπορεί να υποπτεύσει τα κράτη-μέλη. Πώς κάνουν την εφαρμογή του κανονισμού. Τώρα, άλλο. Τι γίνεται με τον ε, έλεγχο, την ανάλυση των ε, πολιτικών μας και της σωματοδικής πολιτικής μας. Γιατί έχουμε κάποιες εκθέσεις για το περιβάλλον, για τη φύση, που περιέχουν αξιόλογα στοιχεία για αυτά τα θέματα. Όμως, θα πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι πολιτικές και πόσο αποτελεσματικές είναι και οι δαπάνες. Πάμε για τη βιωσιμότητα. Υπάρχουν ε, σκόρπιες πληροφορίε αλλά μπορεί η υπηρεσία σας να έχει στοιχεία για τα οικοσυστήματα, για τις πολιτικές προστασίες τους. Και υπάρχει τέτοιου ανάλυση και έλεγχο των περιβαλλοντικών πολιτικών που ασκούνται τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να σας έχουμε εδώ. Μεταξύ είναι σχετικά δύσκολο να υλοποιηθούν σωστές ε, πολιτικές. Η ερώτησή μου είναι ότι αν κοίταξει κανείς τον κατάλογο που μας υποβάλλατε, παραδείγματο χάρη την οδηγία ΝΕΚ, είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν οι πολιτικές αυτές. Είμαστε μακριά ακόμα από αυτούς τους στόχους. Η οδηγία για τις εκπομπές. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση για τις ε, μονάδες καύσης παραδείγματος χάρη, οι στόχοι για, μέχρι το 2020 και μετά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε επίσης πόσο δύσκολο να ελοπιθεί η πολιτική που αφορά τα απόβλητα. Πολλά θέματα λοιπόν και για μένα ένα από τα σημαντικότερα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί έτσι ώστε η συζήτηση για το περιβάλλον να μην είναι ένα είδος ε, χόμπι για κάποιους πράσινους, αλλά να βρίσκεται στην καρδιά για κάθε πολιτική που υλοποιούμε. Γίνει δηλαδή ο αέρας, το νερό, το έδαφος καθαρότερο και να μπορέσουμε να το αφήσουμε σε καλύτερη κατάσταση στα παιδιά μας. Για μένα αυτό θα πρέπει να είναι η καρδιά της πολιτικής μας. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη πόσο μακριά είναι όμως από τις ε, σημερινές ε, προτάσεις. Μπορείτε να μας πείτε πώς το δίκτυο που υπάρχει και λειτουργεί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε αυτές τις πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Γιατί από τη στιγμή που μιλάμε συνολικά στην Ευρώπη για θέματα βελτίωσης του περιβάλλοντος χωρίς το θέμα αυτό να είναι στην ημερήσια διάταξη των Εθνικών Κοινοβουλίων, νομίζω ότι δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Μάλλον λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Εσείς τι προτάσεις έχετε ή εσείς και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την εργασία μας και την αποτελεσματικότητά μας. Αλλιώς κάθε χρόνο θα επαναρχόμαστε και θα ε, μιλάμε για την ε, κακή κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, παρουσίαση. Η σημασία της εργασίας που κάνετε, της ομάδας σας, είναι προφανής. Συμφωνώ απολύτως με όλους όσους σας είπαν ότι χρειαζόσαστε περισσότερα μέσα για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στο μέγεθος της πρόκλησης που έχετε να αντιμετωπίσετε. Mm. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Σήμερα στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει νέος πρόεδρος με διαφορετική άποψη και στάση όσον αφορά το περιβάλλον. Η κατάσταση λοιπόν προφανώς είναι διαφορετική. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τους ε, Αμερικανούς στο πλευρό μας όσον αφορά την υλοποίηση των ε, συμφωνηθέντων και των δεσμεύσεών τους. Ήδη υπάρχουν προσφυγές στα Αμερικανικά δικαστήρια για τις προσπάθειες του νέου Προέδρου όσον αφορετικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όσον αφορά τις ε, βρώμικες μονάδες Υπάρχουν σήμερα και στα ορυχεία κάποιοι εργαζόμενοι που έχουν προσυπογράψει αυτές τις νέες αποφάσεις, τα νέα μέτρα για να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους. Και βεβαίως πάντα το επιχείρημα είναι ότι έτσι θα σωθούν κάποιες θέσεις απασχόλησης. Αυτό όμως δεν είναι μακροπρόθεσμος στόχος ο πλανήτης μας υπερθερμαίνεται και θα πρέπει να δούμε λίγο πιο μακριά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Τι θα κάνουμε για να παραμείνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο πλευρό μας, τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός σας, τι επαφές έχετε με τους συναδέλφους σας ε, στην Αμερική. Δεν βλέπω κάποιον άλλον ομιλητή. Ο κύριος Καπούτο μου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την πρόσφατη έκθεση της ε, υπηρεσίας που μίλαγε για τις ανιώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους του 20. Αλλά, εντάξει, τρία χρόνια μόνο μας μένουν Τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα προσπαθήσει και έχουμε κάποιους ε, τομείς οι οποίοι καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια. Οπότε θα πρέπει να πασχίσουμε να δούμε πώς θα ανοίξουν κάποιες τεχνολογίες με συγκεκριμένο τρόπο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε παγκόσμιο ελληνικές για τους στόχους. Και το είπαμε στην ε, Ρώμη, όπου στη Ρώμη δεν είχαμε κάποια κοινή διακήρυξη γιατί διαφωνούσε η κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Άρα θα πρέπει να δούμε τι πώς θα γίνεται η αποθήκευση, αποθυματοποίηση πορεία με αποτελεσματικό τρόπο όσον αφορά το διοξίδιο Ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδρομή αυτή, αλλά κατά μυστηριώδη τρόπο υπάρχει κάποιο είδου υποτίμηση του προβλήματος της πολιτικής μας. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις προχωρημένε τεχνολογίε που ακόμα δεν υπάρχουν. Εσείς Διευθυντά. Τι λέτε, πώς το βλέπετε. Γιατί αυτά τα θέματα νομίζω ότι είναι τα πιο κρίσιμα τώρα σε αυτή την καμπή της εξέλιξης της ενεργειακής πολιτικής. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Να δώσουμε τον λόγο συντόμως τώρα στους εκπροσώπους του Διευθυντικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας. Ο κύριος Μάικλ Σκούλος Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, δηλαδή να έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα. Μόνο θετικά έχω να πω για το έργο της υπηρεσίας. Είναι μεγάλου βελληνικούς η εργασία αυτή και η σωστή διαχείριση που γίνεται. Ό,τι έχω να σας πω πάντως, για να κάνει και με αυτά που συζητήσαμε, γιατί η υπηρεσία αποτελεί πηγή γνώσης. Πρωτογενός. Όμως θα πρέπει αυτή η γνώση ο κατάλληλος διάβολος να φτάνει εκεί που πρέπει και στην παιδεία και εκπαίδευση. Και αυτό είναι από τα θέματα τα οποία ε, από κάποιο βουλευτή. Μας έχετε δώσει την εντολή να υπενθυμίζουμε στην υπηρεσία για το πώς, ποιοι, ποια είναι τα θύματα των περικοπών. Άρα γι' αυτό και χρειάζεται άμεση σύνδεση με την εκπαίδευση. Επίσης, αυτό το οποίο αναφέρατε, δηλαδή τα προβλήματα που έχουν σχέση με το προσφυγικό σήμερα. Οπότε, αυτά ήθελα να σας επισημάνω. γιατί ίσως όλα αυτά τα παραλάβουμε στα πλαίσια συζήτηση για το πολίτες πρόγραμμα, αλλά δεν βλέπω και πολλές ευκαιρίες όλα αυτά τώρα να εντάσσονται. Και ίσως με την αξιολόγηση της, υπηρε... η εντολή και η σημασία αυτών των θεμάτων ίσως είναι τέτοια που θα ληφθεί τελικά υπόψη. Και κατακλείδη να σας πω ότι ακόμα χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη συμβολή από το ρίζον 2020 και από τα σχέδια τα ερευνητικά. Τα πέρασμα της έλληνας τα οποία σχετίζονται με το έργο μας. Ακόμα δεν υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα τα οποία είναι άσχετα με την ποιότητα της ε, διαχείρισης και διοίκησης της υπηρεσίας, αλλά είναι θέματα τα οποία τα έχετε φύξει στο παρελθόν και εμείς τα έχουμε θέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω όμως πρέπει να το επαναλάβουμε πάλι. Ευχαριστούμε λέει Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καταρχήν, να εκφράσω την εκτίμησή μου για την εξαιρετική εργασία που κάνει ο οργανισμός ε, υπό την προεδρία του Hans Σπρινβίκ. Επί τρία χρόνια ήμουν μέσα του διοικητικό Συμβουλίου και πραγματικά πρόκειται για το πολύ επικοδομητικό κομμάτι αυτής της ευρωπαϊκής συνεργασίας όλους τους ε, εταίρους. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που έτσι και με τον Μάγκλης ε, Βούλης έχουμε υποβάλει στα σχόλια για την περίοδο 2017-2019. Θέμα του περιβάλλοντος και της προστασίας του περιβάλλοντος μας ε, οδηγεί σήμερα σε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από την εποχή που ιδρύθηκε ο οργανισμός. Σήμερα πρέπει πραγματικά να κατανοήσουμε συστημικά και μακροπόθεσμα το περιβάλλον, τη σχέση μεταξύ της ε, κυκλικής οικονομίας, της πράσινης οικονομίας, της οικονομίας σε χαμηλή περιεκτικότητα του άνθρακα και του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος πολλές φορές αντιμετωπίζεται σαν μια πολιτική που απλώς ελέγχει και περιορίζει τον κίνδυνο. Σήμερα υπάρχουν ε, όμως, και αυτό είναι γνωστό σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες και αυτό φέρεται και από τη Συμφωνία του Παρισιού. Χρειάζονται νέοι στόχοι, μακροπρόθεσμοι στόχοι για την μείωση της περιεκτικότητας του άνθρακα, νέοι στόχοι, έγκαιρη πληροφόρηση για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική. Και αυτός μπορεί και πρέπει να είναι ο στόχος αυτού του οργανισμού της υπηρεσίας και η νέα πολιτική της για το μέλλον συνεργασία με την Κίνα για θέματα περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνει πιο σημαντική και να μην βασιζόμαστε μόνο στις νέες πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Να προτείνουμε νέες ε, δυνατότητες ανάπτυξης στην κυβέρνηση της Κίνας πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο ήδη είναι ισχυρό. Βεβαίως εδώ τίθεται και το ερώτημα της διεύρυνσης της εντολής του οργανισμού και των δυνατοτήτων που διαθέτει η υπηρεσία. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καπάντη και τον Μάικλ Σκούλης. Πρέπει να στηρίξουμε σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος την εργασία της υπηρεσίας, να στηρίξουμε ενδεχόμενη αύξηση των μέσων που διαθέτει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς σε μια αποτελεσματική και επιτυχή πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε και εκπρόσωπο από την Κομισιόν, η κυρία Φουσκόντ. Θέλετε να πάρετε το λόγο, εν συντομία. Γεια σας. Δύο λόγια για την αξιολόγηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Επιτροπή σας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ε, και η υπηρεσία. Η διαδικασία ξεκίνησε τον περσμό Δεκέμβρη. Έχουμε μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία συμβουλών η οποία μας βοηθάει να αξιολογήσουμε την ε, ε, υπηρεσία και το IONET. Ε, η εξελόγηση αφορά την περίοδο 2013 μέχρι πέρσι. Είμαστε σε στενή επαφή με την υπηρεσία, την ενημερώνουμε. Η εταιρεία σύμβουλων θα έρθει σε επαφή και με εσάς, ε, ατομικά και συλλογικά, καθώς επίσης και με το κοινό. Η αξιολόγηση θα ε, λάβει χώρα μέχρι το Δεκέμβρη. Μια ενδιάμεση έκθεση θα υποβληθεί γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και θα διοργανώσουμε και ένα σεμινάριο σε συνδυασμό με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Δεκέμβρη. Οπότε αρχές του επόμενου έτους ελπίζουμε θα έχουμε ένα έγγραφο εργασίας με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης τι λειτουργεί καλά, τι χρειάζεται βελτίωση κλπ. Επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης θα σκεφτούμε αν πρέπει να αλλάξει η εντολή, η διακυβέρνηση της ε, ε, υπηρεσίας περιβάλλοντος. αυτή τη στιγμή είμαστε απόλυτα ευέλικτοι, ανοιχτοί συλλέγουμε πληροφορίες. Ευχαριστώ. So, a lot of interest in the... Πολύ ενδιαφέρον και πολύ στήριξη στο έργο της υπηρεσίας σας. Κύριε Μπρένινγκς, τι θέλετε να σχολιάσετε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια, για τις ερωτήσεις και για την ευρεία υποστήριξη που λάβαμε. Αυτό αφορά και την Κομισιόν. Με την Κομισιόν συνεργαζόμαστε πολύ επικοδομητικά. Και παίρνουμε στα σοβαρά τις ε, συστάσεις της. Μίλησα για τους πόρους που διαθέτουμε. Να σας πω ότι το πολιετές πρόγραμμα εργασίας μας είναι μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα γνώσης που στηρίζει τις πολιτικές μας. Οπότε στηρίζουμε την, το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό που έχουμε δει διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν είναι ότι παλιότερα με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο κάθε φορά που μας ε, ανέθεταν ένα έργο ε, μας ε, έδιναν περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα πόστα δηλαδή και μεγαλύτερο προπολογισμό. Τώρα πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε αυτές τις αυξήσεις και πάλι δεν τα καταφέρνουμε. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι πρέπει να είμαστε ορθολογικοί σε ό,τι αφορά τους ε, πόρους που διαθέτουμε. Δεν πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα συναισθηματικά με το θυμικό μας είναι μια λογική, ορθολογική συζήτηση. Αν η Κομισιόν θέλει ποιότητα, εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα ορθολογικό υπολογισμό του τι χρειαζόμαστε. Αυτό ισχύει και έχουμε ότι χρειαζόμαστε για ένα περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων. Όμως, όπως λέμε και εμείς, το λίπος έχει εξαφανιστεί πια και έχουμε φτάσει στους μυς και στα κόκαλα. Εγώ το αντιμετωπίζω ψύχρεμα και προσφέρουμε όσα μπορούμε με καλή ποιότητα. Είπατε, α, υπογραμμίσατε διάφορα θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να εργαστούμε. Να εργαστούμε ενώ όχι μόνο τεχνολογικά ή με συλλογή γνώσης, αλλά πολύ πιο δραστήρια στις δράσεις, να συνεισφέρουμε στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θανάσιο περιβάλλον, για την ε, ατζέντα του Παρισιού, για την ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλα αυτά απαιτούν και τη δική μας συνεισφορά. Σε ό,τι αφορά τις ε, πολιτικές μετάβασεις, νομίζω ότι χρειάζεστε γνώση αλλά χρειάζεται και μια μετάβαση στη γνώση σας. Και αυτό χρειάζεται γνώση και επενδύσεις. Προσπάθησα να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις σας. Μία ε, ομάδα ερωτήσεων αφορά τη διεθνή συνεργασία με τις ΗΠΑ, την Κίνα, ένα κόσμο που αλλάζει ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια πολύχρονη συνεργασία. Έχουμε συνεργαστεί με την υπηρεσία περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Πολλές φορές το χρόνο συνεργαζόμαστε μέσω δορυφορικής κάλυψης, μέσω ε, τηλεσυνεδριάσεων. Ε, ο καινούς διευθυντής όταν λαβέ ανέλαβε τα καθήκοντά του, εγώ ήμουν παρόν και μου είπαν παρακαλώ πολύ ε, ελάτε και ξαναελάτε γιατί μπορεί εμείς να μην μπορούμε να ταξιδεύουμε σε εσά συχνά μπορεί να μας δώσουν, να μας δίνουν την άδεια οπότε επιζητούν αυτή τη συνεργασία από μας και θα το κάνουμε, θα το πράξουμε Είμαστε επίσης σε επαφή με σημαντικά Ινστιτούτα, τεχνολογικά και ερευνητικά Ινστιτούτα των, των ΗΠΑ. Είναι ε, από τα καλύτερα στον κόσμο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα τους, είμαστε σε επαφή μαζί τους και τους συναντάμε στα διεθνή φόρα. Το ίδιο μέρη ισχύει για την Κίνα και, με, και για άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για το έργο μας. Πολύ συχνά όταν δημοσίως πρέπει να προασπίσω το ευρωπαϊκό όραμα, ε, από τη δική μου πλευρά είναι αρκετά εύκολο. Γιατί με 39 χώρες στην υπηρεσία και με 28 χώρες για τις οποίες υφίστανται δεσμευτικοί νόμοι, ε, κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Η ναύτα, η ε, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών της Βορρή Αμερικής έχει ελάχιστε ανταλλαγέ Στην Ασία σχεδόν μηδενικέ. Εμείς είμαστε το μόνο σημείο του πλανήτη που 28 χώρες συν 11 συνεργαζόμενες ε, συνεργάζονται, ε, δουλεύουν μαζί για να δημιουργήσουν δίκτυο γνώσης, για να οργανωθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις, πληροφορίες και βέβαια να επεξεργαστούν δεσμευτική νομοθεσία. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Κίνας αναγνώρισε τα τεράστια προβλήματα που έχει η Κίνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα αυτή τη τεράστια χώρα και μα ρωτούσε εσεί πώ τα καταφέρνετε με τόσο κόσμο, τόσε χώρε. Ε, δυσκολευόμαστε βέβαια να συνεχίσουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά το κάνουμε προ το παρόν. Μόλιση του ατμοσφαιρικού αέρα και σύνδεσή της με την δημόσια υγεία και τις μεταφορές. η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχει τεράστια επίδραση στην δημόσια υγεία. Γιατί δεν βλέπουμε αυτό το άλμα που χρειαζόμαστε, γιατί ένα μεγάλος, ένας μεγάλος αριθμός των ευρωπαϊκών στόχων δεν συνάδουν με τους στόχους του Παγκόσμιου, του Παγκόσμιου Οργάνωσης Υγείας. Έχουμε να καλύψουμε πολύ περιθώριο, πολύ δρόμο. Φανταστείτε τι μείωση θα βλέπαμε στους 460.000 πρόωρους θανάτου, αν τα καταφέρναμε. Ε, η μείωση της χρήσης του τσεκομών του άνθρακα στις μεταφορές, τρεις τελευταίες εκθέσεις έχουμε. Ε, μία που αφορά τις μεταφορές και το περιβάλλον, τον Δεκέμβρη, μετάβαση προς ε, ε, βιώσιμα συστήματα κινητικότητας, δεύτερη έκθεση για, την, ε, για το e-driving. Τι άλλο χρειαζόμαστε εκτός από τον κινητήρα, υποδομές, φορολογικό σύστημα κλπ. Εκεί κοιτάμε, εξετάζουμε σε βάθος το νορβηγικό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή πάνω από το 1 στα 4 αυτοκίνητα που πολλούνται στην Νορβηγία είναι ηλεκτρικά. Χίλιε φορέ περισσότερο δηλαδή από ό,τι σε ορισμένα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σημαίνει αυτό στην Νορβηγία και όχι στι υπόλοιπε χώρε. Και τρίτον, μια έκθεση για την σύνδεση μεταφορών και ενέργεια. Α φανταστούμε ότι όλοι αρχίζουμε και οδηγούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα από αύριο. Τι θα σημαίνει αυτό για τα συστήματα ενέργειας, για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενέργειας ε, κλπ. κλπ. Τώρα, η, η σχέση με τα ενεργειακά συστήματα, ερώτηση του κ. Καπούτο που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή δυστυχώς, ε, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη συστημική προσέγγιση μπορούμε εύκολα να, λέμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε για τα παιδιά μας, αλλά το 2050 είναι ήδη σήμερα. Δεν είναι τα παιδιά μας. Οποιαδήποτε επένδυση κάνουμε σήμερα ε, για καινούριους, καινούργια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας θα λειτουργούν αυτά τα εργοστάσια και το 2050. η, τα παραδοσιακά συστήματα τεχνολογίας και έρευνας μπορούν να μας φτάσουν μέχρι το 2030, αλλά οι επενδύσεις που κάνουμε τώρα θα πρέπει να φτάσουν μέχρι το 2050. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε τις ε, εκπομπές άνθρακα, ε, οξυδίων του άνθρακα και σε επίπεδο εταιρεία αλλά και σε επίπεδο ε, κρατικό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανθράκωση της οικονομίας ε, η οποία θα μας οδηγήσει σε εξοικονόμηση πολλών πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, η σχέση με την αξιολόγηση, νομίζω ότι η Κλάουδια Φουσκάλ σωστά τα εξήγησε, εξήγησε ποια είναι η κατάσταση. Υφίσταται ένας κανονισμός ηλικίας 25 ετών που δεν αναφέρεται καν στην, στον όρο κλιματική αλλαγή. Ίσως θα ήταν καλό να τον ξαναδούμε. Γνωρίζω ότι η δεδηλωμένη πρόθεση είναι να μην καταργηθεί η υπηρεσία μας, αλλά να προσαρμοστεί στην, στα σχέδιά μας για το μέλλον. Αυτή η προσαρμογή θα γίνει επί τη βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Προφανώς εσείς και η Κομισιόν θα το αναλάβετε. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ είμαι ο αξιολογούμενος. Σας ε, καλό να παίξετε ένα δραστήριο ρόλο, αυτό το ρόλο που προβλέπετε και μπορείτε να παίξετε, ένα επικοδομητικό ρόλο τους επόμενους μήνες. Κάποιες άλλες ερωτήσεις αφορούσαν το εθνικό επίπεδο. Πώς μπορούν όλη αυτή η γνώση να προωθηθεί στα εθνικά κοινοβούλια. Έχουμε αυτή την έκθεση του 2015 τότε είχε δημοσιοποιηθεί σε 31 χώρες και βέβαια ε, είχε σχέση και με το Κοινοβούλιο για τη χάραξη εθνικής πολιτικής, οπότε ε, ακριβώς όπως και εγώ και άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι δώσαμε προτεραιότητα στο να διασυνδεθούμε ε, σε αυτό το επίπεδο εθνικής διακυβέρνησης. Καταλαβαίνετε. Και υπήρχε αυτό το πλαίσιο το οποίο το ονομάζαμε επίσκεψη στη σχετική χώρα, οπότε έτσι ε, θέλαμε να έχουμε επαφή στην με την κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή περιβάλλοντος, με το Εθνικό Κοινοβούλιο, με τα στελέχη κάθε κοινοβουλίου, επίσης όποτε επισκεπτόμαστε χώρες για να διορθώσουμε κάποια εκδήλωση, έχουμε πρώτα σε επαφή και λέμε ερχόμαστε, ε, θα πρέπει να είμαστε όσο πιο σωστοί είναι στη διαχείριση του χρόνου ε, και να υπάρχουν ε, αυτά τα πλαίσια για να γίνουν κάποιες ομιλίες, για να συναντήσουμε τα κατάλληλα στελέχη. Αυτό κάναμε και με το δίκτυο IONET. Κάναμε μια στροφή από το δίκτυο που έδινε τα δεδομένα ε, προς ένα δίκτυο το οποίο γεννά γνώση αλλά και κατανόηση σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό όμως γίνεται και επί παραγγελία. Δηλαδή όταν κάποια χώρα λέει βοηθήστε μας στη δυνατοτήτων, εμείς προθύμως πέφτουμε να βοηθήσουμε. Και εμείς το ίδιο ως προς εσάς όποτε μας ζητείτε βοήθεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη δουλειά σας, οπότε όποτε θέλετε ελεύθερα απευθυνθείτε σε μας και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Άλλωστε έχουμε και γραφεία σε όλα τα κράτη-μέλη ή τέλο πάντων έχουμε εκπροσώπους όλων των κρατών μελών στην υπηρεσία. Άρα όλα αυτά γίνονται. Άλλη ερώτηση αφορούσε την οικονομία. Κύριο Ντεμέσμαγκερ αναφέρθηκε ε, στο θέμα απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση, στο σύνθημα ε, της Αμερικάνικης κυβέρνησης. Είπαμε ότι οι φιλόδεξες πολιτικές έχουν βοηθήσει στον να υπάρξει καινοτομία στην οικονομία για επενδύσεις, για θέσεις απασχόλησης για ανταγωνιστικότητα. Και έχουμε ένα σωρό μελέτες που εξηγούν το πώς λειτουργεί έτσι το πράγμα στην Ευρώπη. Αλλά και όχι μόνο. Πάντως, ακόμα. Με εκπλήσει ότι πολλοί είναι κολλημένοι στο, στις τεχνολογίες του περασμένου αιώνα και ελπίζουν ότι έτσι θα φτιάξουν θέσει απασχόληση. Όχι, θέλουμε καινοτομία και έτσι θα χτίσουμε την οικονομία του 21ου αιώνα που θα μα οδηγήσει σε περισσότερη υγεία, σε καλύτερο περιβάλλον, αλλά και στι θέσει απασχόληση όπω όλοι τι θέλουμε για την Ευρώπη. Τώρα όσον αφορά τη συζήτηση για το περιβάλλον. ψάχνω να βρω τι γίνεται όσον αφορά την οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα, την κυκλική οικονομία, με περιβαλλοντική οικονομία, πώς κανείς μπορεί να εξοικονομήσει τους πόρους, γιατί αυτό είναι βασικό στοιχείο της προβληματικής. Επίσης, με το δικό μας θεματολόγιο θα πρέπει να κινηθούμε και να το έχουμε Ευαγγέλιο όποτε συζητούμε την οικονομία. Όχι, όχι, να μην μας ε, περιθωριοποιούν ότι εσείς ασχοληθείτε με τα ζωάκια και τα φυτά και εμείς θα προχωρήσουμε. Και θα σας ρωτήσουμε όταν πάει καλά η οικονομία, όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο. Όχι, τέτοια θέλουμε να είναι η οικονομία στο μέλλον. Θέλουμε να εμπλακούμε στη διαμόρφωση της οικονομίας του αύριο. Αν μη τι άλλο, κόστος και απόδοση, εάν δεν ληφθεί υπόψη η βιωσιμότητα, πάνε περίπατο. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Έχουμε αυτή την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά τέσσερις βαθμούς είπαμε σαν όριο. Ε, τότε θα αποφύγουμε εάν δεν σεβαστούμε αυτό την υποβάθμιση του ενεργειακού κεφαλαίου των φυσικών πόρων. Γι' αυτό έχει σημασία το περιβάλλον και γι' αυτό θα πρέπει να εμπλακεί όταν γίνεται χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Και Υπήρχε και μια κατηγορία ερωτήσεων που αφορούσε την υλοποίηση. Βεβαίω και γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή όλων αυτών. Σε κάθε έκθεση σας δίνουμε και μια λίστα, ένα κατάλογο κρατών με τους στόχους όπως έχουν τεθεί, με τις ε, διάφορες κατηγορίες θεμάτων, τους τομείς και το τι ακόμα πρέπει να γίνει. Γίνεται δηλαδή μια αξιολόγηση. Ε, μερική αξιολόγηση, ολική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος και συζητούμε από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια, με τους ε, εμπειρογνώμονες σε εθνικό επίπεδο για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να είναι πιο καλή η εφαρμογή. Ιδίω όταν πλησιάζουμε στις προθεσμίες για την ολοκλήρωση. Κοιτούμε τη συμμόρφωση, η μη. Αυτή είναι εξάλλου και η εντολή της Επιτροπής. Εμείς δεν συμμετέχουμε στη συμμόρφωση. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε μια υπηρεσία πρώτης γενιάς, όπως θα έλεγα σήμερα. Δεν αποτελεί δηλαδή τμήμα των αρμοδιοτήτων μας. Και από κοινού με την παρακολούθηση και με την αναφορά που κάνουμε στο τέλος θα πρέπει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους εκπροσώπους των κρατών μελών να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση και σίγουρα αυτό θα μειώσει σημαντικά και το κόστος διότι σήμερα προσφεύγουμε σε εταιρείε συμβούλων για την παρακολούθηση αυτών των εφαρμογών. Πιστεύω ότι μια καλύτερη λοιπόν διαδικασία στο μέλλον θα μειώσει σημαντικά και το κόστος. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Καπούτο. Δεν είστε εδώ. Δεν είναι όμως στην αίθουσα. Να πω ότι είμαι αρκετά αισιόδοξο σε σχέση με το πώς έβλεπα τα πράγματα πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Διότι οι μακροπρόθεσμες αλλαγές που συμβαίνουν σίγουρα μας οδηγούν όλους σε μεγαλύτερη δέσμευση. Τα προγράμματα είναι περίπλοκα, αλλά και οι επιπτώσεις, οι συνέπειες είναι πραγματικά σημαντικά πιο σοβαρές. Θα πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να μην διακόψουμε τις προσπάθειές μας. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα μεταφορών στις αστικές περιοχές που να βασίζεται στις συγκεκριμένες παραμέτρους. Και μέχρι το 2050 η εξάλληψη του άνθρακα από τις μεταφορές είναι απαραίτητη. Και οι επιλογές μας θα πρέπει να βασίζονται σε αυτό το στόχο, σε αυτή την καθοδηγητική σε αυτή την κατευθυντήρια γραμμή, σε αυτή την κατεύθυνση, την οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βασιζόμαστε σε πολιτικές του 19ου αιώνα εν ώψη του 2050. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε την σωστή ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος, ο καθοδηγητικός που μπορεί να παίξει η Ευρώπη. Είμαστε πολύ μπροστά όταν πρόκειται για τον τομέα τον ρυθμιστικό. Είμαστε πολύ μπροστά όταν πρόκειται για τεχνολογία, για γνώση. Έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές σήμερα όταν πρόκειται για μετάβαση στον τομέα των μεταφορών. Σίγουρα γνωρίζουμε και κατανοούμε καλύτερα τα προβλήματα στην Ευρώπη σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και όσον αφορά το τομέα της ενέργειας. Να χρησιμοποιήσουμε τις πιο καθαρές, τις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους ε, οικονομικά, ρυθμιστικά εργαλεία, έτσι ώστε όπως στηρίζουμε σήμερα και τη δράση της Επιτροπής, να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένες ε, πληγές, μάστιγες, μόλυνση του νερού, του περιβάλλοντος, του αέρα, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, χρησιμοποιώντας ε, την Ενεργειακή Ένωση, την κυκλική οικονομία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι μελλοντικέ μας δράσεις να στοχεύουν αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να πάτε σε περισσότερες από τις ερωτήσεις που κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, με πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και με μεγάλη χαρά θα συνεχίσουμε την συνεργασία. Χαίρομαστε ιδιαίτερα για την σημερινή σας ε, παρουσία εδώ, τη συζήτηση που είχαμε για τον ε, τρόπο με τον οποίο απαντήσατε στα σχόλιά μας. Θέλετε να ολοκληρώσετε εσείς. Ξέχασα κάτι. Ξέχασα κάτι σημαντικό. Όσον αφορά την ε, διάδοση, την μετάδοση, την επέκταση αυτών που έχουμε σαν γνώση. Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε προγράμματα κατάρτισης για το περιβάλλον. Μπορούμε όμως να παρέχουμε πληροφορίες που πραγματικά θα είναι κατανοητές στους ειδικού. Επίσης, μπορούμε να συνεισφέρουμε με τα ερευνητικά κέντρα τα πανεπιστημιακά. Εγώ συχνά πάνω από 10 φορές το χρόνο παίρνω το λόγο και κάνω ομιλίες ε, σε πανεπιστημιακά κέντρα και κέντρα έρευνας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε. Θα σε ευχαριστούμε πολύ. So, uh, dear colleagues, uh, this uh, concludes our agenda for today. And... Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Θα ήθελα να σας πω ότι αύριο θα ξεκινήσουμε στις 10.30 με τις ψηφοφορίες και στις 9 θα λάβει χωρίς συνάντηση των συντονιστών.